All right, everybody, if you could take your seats. I know there's a slight seating crisis. Καθίστε, βλέπω πως υπάρχει ένα πρόβλημα στα θεωρία. Only members in members seats and only assistants. Παρακαλώ στις θέσεις των βουλευτών μόνο βουλευτές και στις θέσεις των βοηθών μόνο βοηθή. So if we all sit down, then we can see where να καθίσουμε για να δούμε πού περισσεύει χώρος. Λυπούμε για το ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα, αλλά πάμε να αλλάξει στις διάφορες αίθουσες οι επιτροπές. Οπότε αυτή τη φορά βρεθήκαμε σε μια μικρή αίθουσα με ενδιαφέρον θέμα. Και εγώ υποφέρω. Ο ίσως μου πάει και το βλέπει από το ίντερνετ. Εκτός αν έχει βρει εδώ πέρα καμία θέση. Okay, uh, right. Um, we are now having a hearing on CRD. Περνάμε λοιπόν στην ακρόαση για την οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων υπαριθμών 4. Θα συνεχιστεί μέχρι τι 5.30 το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να σα κάνω εισαγωγή τώρα για την διάσημη αυτή τέταρτη οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων. Είμαστε τυχεροί που ο Ανδρέα Ανδρέα βρίσκεται εδώ πέρα για να μας κάνει μια εισαγωγή από τη σκοπιά του Ευρωπαίου Επόπτη και μετά θα περάσουμε σε ένα πάνελ ενδιαφερομένων τους οποίους θα ακούσουμε με τη σειρά και μετά θα περάσουμε στις ερώτα και τη συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν να είστε σε φόρμα. Λοιπόν, Ανδρέα, χαιρόμαστε που σε ξαναβλέπουμε οπωσδήποτε, θα έχεις ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία από το καλοκαίρι του 2007 αποκάλυψε μεγάλες αδυναμίες στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα μαθήματα τα οποία αντλήσαμε μέχρι στιγμής μας δείχνουν μια ευρεία συνένεση και σύγκληση στο διεθνές επίπεδο στο τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει στο ρυθμιστικό τομέα. Το 2009 στις ε, συστάσεις της για την Ευρωπαϊκή Εποπτεία και Ρύθμιση, η υψηλή ομάδα υπό την Προεδρία του Ζάκ Τελεαροσχέ τόνισε την ανάγκη του να πάμε σε ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, ενισχύοντας τις απαιτήσει για ποιότητα και ποσότητα τραπεζικού κεφαλαίου, να μειωθούν οι προκυκλικές τάσεις, απαιτώντας βεβαίως ε, να υπάρχει ρευστότητα η οποία θα σωρεύεται τους καλούς καιρούς για να είναι ευκαιροί τους χαλεπούς. Η ίδια έμφαση βεβαίως δόθηκε και από τους ηγέτες των G20 στο Pittsburgh το Σεπτέμβριο του 2009 και επιβεβαιώθηκε όταν το νέο διεθνές πλαίσιο στο οποίο συμφώνησε η Επιτροπή της Βασιλείας του 2010 εγκρίθηκε από τους G20 στη Σεούλ τον Νοέμβριο του 2010. Η πρόταση της Κομισιόν του Ιουλίου του 2011 συμφωνεί πλήρω και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται η πρώτη δικαιοδοσία στον κόσμο η οποία φέρνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο. Προετοιμάζοντας λοιπόν αυτό το νέο πλαίσιο είχαμε και την έκθεση του Μακάρας πριν από ένα έτος. Η αρχή μας λοιπόν καλείται να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσω της ε, σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελούν τους ενιαίους κανόνες. Ως μια νέα αρχή μα τιμά το ότι η Κομισιόν μας ανέθεσε αυτέ τι ε, ευθύνε και αναμένουμε την οριστική απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Βεβαίω, ανησυχούμε για το τεράστιο ποσό Τεράστια ποσότητα ευαίσθητη τεχνική δουλειά θα πρέπει να γίνει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ε, διαδικασία του ατύπου διαλόγου, της ε, μελέτης αντικτύπου και τη δημόσια διαβούλευση, αλλά είμαι πεπισμένος μπορούμε να επιτύχουμε αρκεί να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και να βασιστούμε σε αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας, έχοντας βέβαια και την εμπειρία που υπάρχει σε εθνικές εποπτικές αρχές. Οι τεχνικές ε, τεχνικές προδιαγραφές μας θα πρέπει βεβαίω να αποφεύγουν τις σημαντικές αποκλήσεις οι οποίες υπήρχαν στην εθνική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης και έχουν προκαλεί σοβαρή βλάβη πριν από την κρίση, καθώς οδηγούσαν σε νομική αβεβαιότητα, άφηναν το πεδίο ανοιχτό σε διοικητικό ανταγωνισμό για να ωφελήσουν εθνικε, εθνικούς ε, πρωταθλητές και βεβαίως ήταν δύσκολο για τις εταιρείε να, λειτουργήσουν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Ένα από τα βασικά μαθήματα της κρίσης λοιπόν είναι πως η χαλάρωση των ρυθμιστικών κριτηρίων και ο ανταγωνισμός στη χαλαρότητα για τον ορισμό του κεφαλαίου είναι κάτι το οποίο βλάπτει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι η άποψή μας πως μόνο μέσα της υψηλότερης ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Tier 1 των Ίδρυματων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτές τις αυστηρές απαιτήσει με συνεχή παρακολούθηση για να μην υπάρχει μια χαλάρωση της ποιότητας του κεφαλαίου των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Ιδρυμάτων ήδη. Ακολουθούμε αυτή την πρόκληση όταν μιλάμε για τον ορισμό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για τα τελευταία stress test τα οποία είχαμε και ελπίζουμε πως δεν θα αφαιθεί πλέον χώρος για εθνικέ ερμηνείες και θα έχουμε ένα ενιαίο σετ κριτηρίων της υψηλότερης ποιότητας. Οπότε θα υπάρχει ένα κοινό κεφάλαιο όσον αφορά την μονιμότητα, τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών και την ευελιξία στις πληρωμές. Βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινό ορισμός του κοινού κεφαλαίου, οπότε θα πρέπει να μην υπάρχει η δυνατότητα να εξασθενήσουν οι απαιτήσει στο εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κοινή εφαρμογή σε ολόκληρη την κοινή αγορά. Το άρθρο 24 παράγραφος 4 απαιτεί από την αρχή μας να συντάξει και να δημοσιεύσει την ε, αρχή και βεβαίως θα πρέπει να δημοσιεύσουμε και τα μέσα τα οποία θα έχουμε στην διάθεσή μας. Το δεύτερο σημαντικό είναι η αύξηση των κεφαλαίων απαιτήσεων ε, στο πλαίσιο της ε, μόχλευσης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Βεβαίως ε, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο λέει πως έτσι θα εμποδιστούν τράπεζες να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την εμπειρική ανάλυση που έχει γίνει από τις εποπτικές αρχές. Ένα υψηλότερο επίπεδο κεφαλίου θα μειώσει την, δυνατότητα, την πιθανότητα χρεοκοπία των τραπεζών και το κόστος χρηματοδότησης. Αυτές οι μέρες ήδη παρατηρούμε πως ε, εάν δεν θεωρείται πως οι τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες ε, χρηματοδότησης, κάτι το οποίο μπορεί να έχει πιθανότητες απομόχλευσης βεβαίως. Θα πρέπει ο λόγος αυτός να συνδεθεί με έναν λόγο μόχλευσης για να υπάρχει μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τον κίνδυνο. Κάποιοι λένε πως ο λόγος αυτός μόχλευσης θα πρέπει να είναι το μόνο μέσο που έχουν οι εποπτικές αρχές στην διάθεσή τους γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα μέσα μέτρησης. Εγώ θεωρώ πως οι δύο αυτοί λόγοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και οι εποπτικές αρχές να έχουν ένα εργαλείο εξέτασης των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Τρίτον, η εισαγωγή μακροπροληπτικών μέσων θεωρώ πως είναι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες ως απάντηση στην κρίση το νέο πλαίσιο εισάγει έναν, ε, μια αντικυκλική προστασία για να υπάρχει ήδη μια, καθώς και κάποια άλλα μακροπροληπτικά εργαλεία. Οι εθνικές πολιτικές αρχές θα πρέπει να έχουν ε, την ε, ευελιξία να χειρίζονται αυτά τα κεφάλαια και θα πρέπει βεβαίω να έχουν μια διακριτική ευχέρεια. Για να υπάρχει λοιπόν ενιαία αντιμετώπιση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να ε, δώσει κάποιες κατευθύνες γραμμές εξάντε και να κάνει κάποιους ελέγχους εξ Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί κάτι το οποίο συχνά λέει ο κλάδο, πω ε, η απελευθέρωση αυτών των κεφαλαίων σε περίπτωση κρίση θα είναι δύσκολη λόγω τη πίεση των αγορών. Τέταρτον, η πρόταση για την ε, ΟΚΑ 4 θα φέρει ένα αυξημένο κίνδυνο καθώς ε, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Βασιλείας 3 και θα φτάσουμε το επίπεδο κάλυψης της ρευστότητας μέχρι το 2015 και στο 2018 θα έχουμε φτάσει στο σταθερό επίπεδο χρηματοδότησης. Γνωρίζω βεβαίως πως ο κλάδος ανισχύει πάρα πολύ για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων και πιστεύω πως θα πρέπει να αξιολογήσουμε το τυχόν θέλετε συνέπειες κατά τη διάρκεια της περίοδου παρατήρησης. Βεβαίως υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν υψηλά κεφάλαια τα οποία θα είναι διαθέσιμα ακριβώς για να αντέξουν περιόδους ε, στρες και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την, ε, τον μετασχηματισμό τυχών ε, ομολόγων τα οποία λύγουν. Βεβαίως η αρχή μας θα αρχίσει να επιτηρεί και τους δύο αυτούς λόγους, ο οποίους αναφέραμε από το 2013, ιδιαίτερη έμφαση στην ε, επίπτωση που θα έχουν στο δανεισμό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επίση, όπως αναφέρθηκε και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2011 για την οικονομική και κοινωνική κρίση, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και των τριών υποπτικών αρχών είναι ένα βασικό βήμα για να υπάρχουν ενιαίοι κανόνε, αλλά απαιτείται περαιτέρω πρόοδο για να υπάρχει ενιαία εφαρμογή αυτών των κανόνων. Τις ε, τελευταίες δύο δεκαετίες υιοθετήσαμε μια προσέγγιση η οποία εστιάζεται και βασίζεται στην εσωτερική μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων εντός των εταιριών. Το ότι δώσαμε αυτές τις ε, αρμοδιότητες στις υπορρύθμιση εταιρείε είχε βαθμό επιτυχίας ο οποίος διέφερε. Εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά την εποπτεία Άρα θα πρέπει να αναπτύξουμε στιβαρές μεθοδολογίες για την ε, εποπτική λειτουργία και την αξιολόγηση, καθώς και μηχανισμούς αξιολόγησης απομοτήμους για να εφαρμοστούν οι μεθοδολογίες αυτές με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολη αυτή η πρόκληση και δεν θα καταφέρουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Όμω θα πρέπει να υπάρξει σταθερή πρόοδο και η εφαρμογή θα μα δώσει μια νέα ευκαιρία για να προωθήσουμε τη σύγκληση. Βεβαίως το να έχουμε ενιαία ρύθμιση είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που πηγαίνει πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα η Συμφωνία και τη Βασιλεία 3 θα πρέπει να εφαρμοστεί ομοιόμορφα στο παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη η Επιτροπή της ε, Βασιλείας έχει ανακοινώσει πως θα ε, υποβάλει νέες προτάσεις για καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση. Επίσης ε, η πρόταση την οποία έχει υποβάλει η Κομισιόν προσαρμόζει κάποιε παγκόσμιε προδιαγραφέ στι ιδιαιτερότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω παραδείγματο χάρη το επιχειρηματικό μοντέλο Τράπεζα Ασφαλιών, που είναι ένα παράδειγμα όπου διαφέρουν ε, και θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνε τη Βασιλεία. Και άρα θα πρέπει να μην προσφέρουμε εύκολου τρόπου στι τράπεζε να παρακάψουν του αυστηρού κανόνε κεφαλαιακή επάρκεια. Επίση, Αυτά δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τι τράπεζε οι οποίε δραστηριοποιούνται διεθνώ, αλλά για όλε τι τράπεζε και επενδυτικέ εταιρείε που έχουν άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ευρύ πεδίο εφαρμογή απαιτεί να δώσουμε την σωστή έμφαση στην αναλογικότητα για να λάβουμε υπόψη του ιδιαίτερου κινδύνου τη κάθε τράπεζα και την διαφοροποίηση που υπάρχει στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον κάθε αυτό συμφέρον στο να εφαρμόσει τι νέε αυτέ ε, προδιαγραφέ για να αυξηθεί η αντοχή του τραπεζικού συστήματο, όμω η αποτελεσματικότητα τη εφαρμογή θα μπορούσε να υπονομευθεί εάν δεν γίνουν αυτά ταυτόχρονα ή με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό είμαστε σε έναν διάλογο με την Κομισιόν και τι τρει ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Thank you very much. Uh, uh, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατήσατε και το χρόνο Οπότε τώρα ερχόμαστε στους ενδιαφερομένους ε, φορείς. Θα λάβετε το λόγο με τη σειρά που είσαστε εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα. Ντομινίκ Γκραμπέρ λοιπόν, πρώτα απ' όλα από την BNP ε, Paribas που είναι η συνεκεφαλής ε, των δημόσιων και πολιτικών υποθέσεων του ομίλου. Θέλω να ευχαριστήσω που, τον κύριο Καράς που μας κάλεσε και να σας ε, ευχαριστήσω που μας δείτε τη δυνατότητα να λάβουμε το λόγο. Θα σας παρουσιάσω τη μαρτυρία μιας ε, τράπεζας η οποία έχει επιλέξει, έχει στιγματίσει πέρα της Ευρώπης, ε, δραστηριοποιείται σε τέσσερις αγορές εντός Ένωσης, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, πάνω από το 5% του κεφαλαίου της είναι η λιανική τραπεζική δραστηριότητα, ένα τρίτο δραστηριότητα είναι η ε, τράπεζα χρηματοδότησης επένδυσης για τη χρηματοδότηση κρατών ε, επιχειρήσεων και διαχείριση κινδύνων των πελατών. Όχι όμως δραστηριότητα συναλλακτική, trading ε, ίδια. Και το ένα έξι, το έκτο Πρόκειται για επαγγέλματα διαχείρισης αποταμιεύσεων. Έχουμε λοιπόν διαφοροποιημένο πρόγραμμα και γεωγραφικά και έτσι καταφέραμε χωρί να αστοιχήσει η κρίση στου Γάλλου φορολογούμενου να ξεπεράσουμε βρόχης πώ τα εμπόδια. Θέλουμε να ε, καλωσορίσουμε την έγκριση του πακέτου Βασιλεία 3 από την Κομισιόν ε, και βέβαια ε, διατηρείται και το πλαίσιο της, το πνεύμα μάλλον της Βασιλείας, διότι η κυριαρχία της ε, τραπεζικής διαμεσολάβηση στην Ευρώπη, η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών μοντέλων και η ανάγκη διατήρηση, του, η επιθυμία διατηρήσή του είναι λόγια που ε, δικαιολογούν τι ε, διαφορές που μπορεί να υπάρχουν με το κείμενο της βασιλεία, Μιλάω για την ΟΚΑ 4. Πιστεύουμε πάντως ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο μας να διαχειριστούμε τις κρίσεις και η Ευρώπη θα μπορέσει να ε, είναι ένας παγκόσμιος ε, παίκτη. Μία πρώτη παρατήρηση για τη Βασιλεία Τρία θα εφαρμοστεί ε, προληπτικά. Οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες πρέπει να φτάσουν έναν στόχο κεφαλαίου ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2013 έξι έτη δηλαδή πριν το στόχο που ορίζεται στον κανονισμό. Οι γαλλικές τράπεζες και οι ελβετικές τράπεζες θα μπορούσατε λίγο να ε, επιβραδύνετε, πηγαίνετε πάρα πολύ γρήγορα και διαβάζετε κιόλας. listening in English to the interpreter, so um, if you want if you want us to understand, slow down. Αν θέλετε να γίνετε κατανοητοί, παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά. Λοιπόν, οι γαλλικές και ελβετικές ε, τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα σεβαστούν ε, το σύνολο των κεφαλαιακών κανόνων από την 1η Ιανουαρίου 2013 δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις, κεφαλακές απαιτήσεις είναι την εφαρμογή όλων των, αφε, των μειώσεων και εκτόσεων. και η σταδιακή ε, υλοποίηση ξεκινάει από το 2014 και έχουμε και την αύξηση των σταθμισμένων ε, στοιχείων των ενεργητικού Δηλαδή, ο K3 είναι κίνδυνος ανταλλάγματος ε, στις ε, πράξεις που προβλέπονται από το κείμενο της Βασιλείας 3 δεν αποκλείεται και άλλες ε, τράπεζες λόγω των αγορών αναγκαστούν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Αυτό πολύ συγκεκριμένα μεταφράζεται από τις πρώτες αναγγελίες μειώσεων ε, ένας από τους στόχους άλλωστε των εποπτών. Σε ό,τι αφορά τις γαλλικές τράπεζες ε, θα μειώσουν ε, κατά 10-15% τις δραστηριότητες εμπορικής τράπεζας και τράπεζας χρηματοδότησης. Εκεί δηλαδή που ήταν ηγετικές όπως η χρηματοδότηση αεροναυπηγικής ή αεροναυπηγικής βιομηχανίας, αυτή η θέση θα καταληφθεί από ξένες εταιρείες, Ιαπωνία, από αμερικανικές ή κινέζικες. Αυτό βέβαια είναι και η ουσία του ανταγωνισμού, θα μπορούσε να πει κανεί, αλλά είναι και το μοντέλο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών τραπεζών που ακολουθούν τη διεθνή ανάπτυξη των πελατών. Αυτό το μοντέλο τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ίσως τελικά ε, πιο πολλά Boeing παρά Airbus θα παίρνουν αυτή τη χρηματοδότηση. Τώρα, αναπτύχθηκε η Βασιλεία 2 γιατί η Βασιλεία 1 παρότρινε στην ανάληψη κινδύνων. Και για την ίδια στάθμιση κεφαλαίου οι τράπεζες έχουν συμφέρον να αναλάβουν το μέγιστο κίνδυνο για να έχουν και τη μέγιστη αποδοτικότητα. Ενώ στη Βασιλεία 2 έχουμε ένα προληπτικό ε, καθεστώς ε, που είναι ευαίσθητο στους κινδύνους. Ε, οι συζητήσεις ακριβώς για αυτά τα σταθμισμένα στοιχεία εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παρουσιάζουν ε, σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού που είναι πιο μικρά σε σχέση με τις αμερικανικές τράπεζες γιατί δεν έχουν τόσο ε, μεγάλο ποσοστό κινδύνου στους ισολογισμούς τους. Στην Αμερική έχουμε πολύ μεγάλη τιτλοποίηση. 6,5 φορές περισσότερη το 2006 στη ΣΥΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη 11 τράπεζε του χρόνου λοιπόν θα περάσουν στο, στη Βασιλεία 2. Ε, η επικύρωση των μοντέλων γίνεται στο εσωτερικό επίπεδο. Υπάρχουν οι ανάλογε υπηρεσίε αξιολόγηση των κινδύνων, ανεξάρτητα από τον εμπορικό τομέα. Και στη συνέχεια εγκρίνονται από του επόπτε. Υποβάλλονται στο backtesting σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, δηλαδή, ε, βλέπουμε τι ελαττώματα υπήρχαν και αυτά συγκρίνονται με τα ε, προβλεφθέντα. Και υπάρχει ένα ακόμα στρώμα προστατευτισμού το οποίο Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία των εσωτερικών μοντέλων. Έχουμε κάποιες, ε, κάποια προβλήματα ε, και με τα εσωτερικά μοντέλα ε, και με τα μοντέλα των εποπτών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν θετικά. λόγος μόχλευσης ε, ουσιαστικά είναι ένα απομεινάρι του, της Βασιλείας 2. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει στον δεύτερο πυλώνα, γιατί θα μπορούσε αν έμπαινε στον πρώτο πυλώνα, να αποθαρρύνει τους επενδυτές και τους επόπτες να προβούν σε αναλύσεις κινδύνου, όπως είναι η ταξινόμηση ΑΑΑ των δομημένων προϊόντων και αυτό ε, δεν θα ε, οδηγούσε στη θέουσα επιμέλεια τους ε, επενδυτές. ο δείκτης ρευστότητας και οι αδυναμίες του έχουν εντοπιστεί στην πρώτη έκθεση καράς και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της κρίσης του δημόσιου χρέους. Θα πρέπει λοιπόν αυτόν τον λόγο να τον ελέγξουμε και να τον δοκιμάσουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα QIS της Βασιλείας δεν λαμβάνουν υπόψη το template της ΟΚΑ 4 και οι οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να εκτιμηθούν σε ένα πλαίσιο μεγάλης δημοσιονομικής εξυγίανσης και στενών περιθωρίων ελιγμών. Έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η περίοδος παρατήρησης ε, θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη, τον απαιτούμενο λόγο ρευστότητα, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να οριστούν ποιοι θα είναι οι παρατηρητές, ε, θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκεί εκπρόσωποι των πελατών των τραπεζών, των επιχειρήσεων, των ε, ΜΜΕ, των ε, ε, πελατών λιανικής πόλης, εκπροσώπων κεντρικών τραπεζών κτλ. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν την επικύρωση των συλλαγέντων δεδομένων και την ανάλυσή τους, καθώς και την εκτίμηση των προσδοκόμενων αλλά και μη προσδοκόμενων επιπτώσεων των κανόνων υπολογισμού στις οικονομίες. Έπειτα θα πρέπει ε, να έχουμε μια ποιοτική διαδικασία ανάλυση των αλλαγών, ε, να δούμε δηλαδή, χωρίς βέβαια κανένα, ε, καμία προκατάληψη, των κλάδο και τι αλλαγές προκύπτουν. Σίγουρα θα γίνουν πολύ σημαντικές ανακατατάξεις, διότι υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο originate to distribute Καλό θα ήταν λοιπόν να καταλάβουμε όλες αυτές τις αλλαγές και μετά να υλοποιηθούν. Επίσης θα πρέπει να οργανωθεί αυτή η μετάβαση σε ένα πλαίσιο χαμηλής ανάπτυξης. Θα αναλυθούν μια σειρά από ζητήματα, σε ό,τι αφορά τα ε, ρευστά στοιχεία ενεργητικού, βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν ε, μη ε, ρευστά ακόμα και στην ζώνη του ευρώ τα χρέη, τα δημόσια χρέη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη διαφοροποίηση αυτής της, ε, του μηχανισμού προστασίας ρευστότητας. Τώρα, επιπτώσεις στη μακροοικονομική χρηματοδότηση γιατί θα μπορούσαν να υπάρξουν αναταράξεις στην ε, χρηματοδότηση. Έχουμε επίση ε, τα δάνεια στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη χρηματοδότηση των υποδομών, των εξαγωγών ε, διαφόρων έργων ε, του διεθνούς εμπορίου. Όλα αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει να διαδραματίσει τη διαδικασία αυτή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτή η περίοδος παρατήρηση το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορέσει να προλάβει κάποιες εξέλιξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, γι' αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο συναπόφασης. Εν κατακλείδη, ο K4 ήδη έχει αποτελέσματα πρωτού καν εφαρμοστεί. Θα υπάρξουν μειώσεις ε, στη χρηματοδότηση. Δεν επιτυχάνεται κατά την άποψή μας πλήρως ο στόχος της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, Αυτό θα εφαρμοστεί πολύ λίγο στη ΣΥΠΑ που είναι και η πηγή αυτής της κρίσης. Άρα για να αποφύγουμε ε, το συστημικό κίνδυνο, νομίζω ότι καλό είναι να επιτρέπουμε την ελεγχόμενη χρεοκοπία στις ε, τράπεζες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε αμέσως στον Άντρα Σερτάξερ, που είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, αντίστοιχης τράπεζας. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά να μπορώ να σας προσφωνήσω και πάλι, αλλά αυτή τη φορά για το κρατικό χρέος, την κρατική υπερχρέωση. Για το ίδιο θέμα που είχα προσκληθεί να παρέμβω δύο χρόνια πριν, όταν είχαμε τη χρηματοοικονομική κρίση. Στο μεσοδιάστημα όμως έχουμε τη Βασιλεία 3 και τη μεταμόρφωση της ε, Βασιλείας 4 στο CD4 ε, ε, που έχουμε προχωρήσει. Γενικά τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν δράση ώστε να αποδεχθούν αυτοί, αυτές τις κινήσεις και το βρίσκουν ένα θετικό ε, έγγραφο. Αναλογίες κεφαλαίων που είχαν αμφισβητηθεί στο παρελθόν τώρα θεωρούνται κάτι το φυσικό. Ποσοστά ρευστότητα που πριν από δύο χρόνια έλεγαν όλοι είναι αδύνατο να φτάσουμε εκεί, είναι τώρα κάτι το εφικτό. Το πρόβλημα που βλέπουμε είναι ότι δεν πρόκειται να είναι ισότιμο πεδίο δράσης ε, για όλους τους εμπλεκόμενους στην Ευρώπη. Διότι πολλές χώρες ε, στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει τις επιδιαιτησίες για τη Βασιλεία Τρία και απαιτούν ακόμα υψηλότερα κεφάλαια. Ακόμα και στις Βρυξέλλες έχουμε συζητήσεις ε, για αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Εργάζομαι για μια τράπεζα που έχει που έχει, κάνει μια, έχει λάβει μια πολύ σημαντική απόφαση, εχθές κιόλα. Και τι είναι αυτή. Αυτή είναι ότι για μας έχει αλλάξει πλέον ο κόσμος και άρδιν δραματικά. Και μάθαμε κάτι επώδυνα, με επώδυνο τρόπο, ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο. Δανείσαμε υπερβολικά πολλά ποσά, μεγάλα ποσά, σε πάρα πολλούς δανειστές και κυβερνήσεις που δεν άντεχαν και δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιο βάρος δανεισμού σε τέτοιο μεγάλο όγκο. Κάνουμε λόγο για την η υλοποίηση του ε, CRD4 και απαιτούνται οι τράπεζες πλέον να αυξήσουν τα κεφαλαία τους, την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε χρονική περίοδο που η κατάσταση του κρατικού χρέους σε πολλές από τις ευρωπαϊκές ε, χώρες δεν έχει επιληθεί, δεν έχει αντιμετωπιστεί καθόλου. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πορευόμαστε στην Ευρώπη προς μια ακολουθούμε μια πολύ επικίνδυνη πορεία διότι αν είναι κάποιος τράπεζα σε μια χώρα και λειτουργεί έτσι, σε μια χώρα που δεν παίρνει ιδιωτικά κεφάλαια και χρηματοδότηση πλέον, και αν έχει κανείς ποσόστοση κεφαλαιακή, οποιαδήποτε και να είναι, 8%, 10%, 12% ή 15% ή 18% είναι τελείως άσχετο και αδιάφορο αν έχει κανείς πολλά ομόλογα μια τέτοιας χώρας ως χρέος της και δεν υπάρχει ιδιωτική κεφαλαιοδότηση, πάει, τελείωσε, χρεοκόπησε κανείς, χρεοκόπησε κάποιος. Έτσι λοιπόν η επίλυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών χωρίς να επιληθεί το ευρωπαϊκό πρόβλημα υπερχρέωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει με κανένα τρόπο αποσυνδεδεμένα. Γι' αυτό αποφασίσαμε ως μια μικρή τράπεζα στην κεντρική Ευρώπη ότι, αποφα... ότι δαπανίσαμε υπερβολικά κεφάλαια επενδύοντας σε μια τράπεζα στη Ρουμανία. Δώσαμε υπερβολικά, για παράδειγμα, δάνεια σε πελάτες στην Ουγγαρία και σε σχέση και με τα ε, ελβετικά φράγκα. Ήταν λάθος να, δανείζουμε όσον αφορά και για την προμήθεια CDR, Credit Default Swap, CDS με συγχωρείτε. Και ήταν πράγματι πολύ επώδυνη αυτή η κατάσταση. Αισθάνομαι όμως πολύ καλύτερα σήμερα. Πολύ καλύτερα αισθάνομαι σήμερα, διότι τελειώσαμε πια με αυτά και μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια νέα φετηρία πλέον. Θα έλεγα ότι η δουλειά για το, την Βασιλεία 3 και εγώ δεν ήμουν πολύ υπέρ της Συμφωνίας Βασιλείας 3 στην αρχή. Τώρα την εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι πολύ αξιόλογο έργο αυτό. Και όσον αφορά το έργο στο ε, CRD4, ε, Capital Requirements Directive 4, είναι πολύ καλά. Μόνο που προσπαθούν κάποιοι να αλλάξουν τα πράγματα μόνοι τους. Γιατί δεν δεχόμαστε τη Βασιλεία 3 ως έχει, χωρίς αλλαγές. Είναι τέλεια και θα κάνει τις εργασίες των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων των τραπεζών πολύ καλύτερη. Πολύ, θα λειτουργούν όλα πολύ καλύτερα. Τώρα και με την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων όσον αφορά τον δανεισμό της ε, στην πραγματική οικονομία οι υψηλή συχνότητα οικονομικές συναλλαγές έχουν αστεί το τελευταίο καιρό και δεν θα πρέπει λοιπόν να, ακολουθήσουμε μια πορεία συρρήκνωση. Αν κάνουμε λόγο για αυτά τα πράγματα που θα θέλαμε να αλλάξουν και επιτρέψτε μου εδώ έχω μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω και είμαι συναισθηματικά θα έλεγα φορτισμένος για αυτό το θέμα. Και ιδιωτελώ, μια και έχουμε μια τράπεζα στην κεντροανατολική Ευρώπη και δεν έχουμε κεφαλαϊκέ αγορέ. Και εμεί εξαρτώμαστε ακόμα περισσότερο από ό,τι άλλε τράπεζε στην Γερμανία ή στη Γαλλία, απόλυτα από τον τραπεζικό δανεισμό. Και χρειαζόμαστε αυτόν τον τραπεζικό δανεισμό. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Και αν η Συμφωνία Βασιλεία 3 εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο, και έτσι σε σχέση με μη αξιολογημένες, μη συγμένες ή αξιολογημένες εταιρείε ε, ο δανεισμός ε, αν μπορεί να διευκολυνθεί, αυτό που θα κάνουμε είναι τις υποθήκες, τα ενυπόθηκα δάνεια σε ελβετικά φράγκα από την Ουγγαρία θα πρέπει να ε, αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία με το subprime lending στις ΙΠΑ δηλαδή τα δάνεια τα οποία ήταν αναξιόπιστα σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ. Κάναμε λοιπόν, συνήψαμε κακά δάνεια, αρνητικά δάνεια και πληρώνουμε τώρα εμείς. Πληρώνουν οι πελάτες μας, πληρώνουμε και εμείς. Αμφότεροι και οι πελάτες και εμείς ως τράπεζα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες περισσότερες λεπτομέρειες συνάπτουμε αρνητικά δάνεια και τα, και τα φορτωνόμαστε και τα φορτώνονται και άλλοι. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να, να αντιμετωπιστεί αυτό είναι η Βασιλεία 3 και το CDA 4 CRD4 να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο δανεισμού που θα είναι μικρότερο. Το να είναι κανείς μικρός σημαίνει αυτόματα σήμερα ότι είναι κακός. Αν έχουμε όμως μια εταιρεία που δεν έχασε χρήματα τα τελευταία 50 χρόνια, μια εταιρεία που ήταν πελάτης μας για 100 χρόνια με 50% σε ομόλογα και 50% σε ε, αποταμίευση και έτσι δεν είναι δυνατόν ε, να ε, ξεφύγει από τις λαβίδες. Λόγω αυτού είναι αυτόματα κακή μια τέτοια εταιρεία και πρέπει να επιβαρύνονται λοιπόν οι συναλλαγές με αυτήν. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, είναι ακατανόητο, παράλογο και στρεβλό και δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ο δανεισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευκολυνθεί και να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Και ο μόνος τρόπος, το μόνο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι αφορά την αντιμετώπιση των μειονοτήτων όσον αφορά τους μετόχους, γιατί αυτό μας αφορά άμεσα. Καταρχήν είναι μια ευφυής, ένα ευφυές εργαλείο αυτό να μειώνει κανείς τη διαθεσιμότητα ε, των, ε, την, παρέμβαση μειονοτικών συμφερόντων. Ε, όμως θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό σε μια ομάδα τραπεζών παγιωμένη όσον αφορά τις συμβατικές της ε, δραστηριότητες ε, συναλλαγών. Κάθε μία θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη έναντι των οφειλών των, της άλλης, όπου κάθε μικρή τράπεζα η οποία ε, συνεργάζεται ή συναρτάται με μια άλλη θα ε, επιβαρύνεται και θα δεσμεύεται όσον αφορά τις υποχρεώσεις άλλης. Θα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αν μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοιου είδους εξαίρεση, διότι το σύστημα των ε, αποταμιευτικών τραπεζών είναι πολύ θετικό. Μπορεί να εξυπηρετεί τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις στα χωριά τους, επιτόπου. Πολύ καλύτερα από ό,τι μπορούν να το κάνουν οι μεγάλες τράπεζες. Είναι ένα πολύ καλό σύστημα να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί η σταθερότητα, του ε, χρηματοπιστωτικού μας συστήματος στην Αυστρία, στην Κεντρική Ευρώπη. Αν κάτι θα μπορούσε να γίνει υπέρ αυτής της κατεύθυνσης θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, and... ευχαριστώ πολύ. Επόμενη είναι η Κλάουντια Μπούχ, προκαθηγήτρια διεθνών μακροοικονομικών ε, και οικονομικών, επιστημονική διευθύντρια στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία μου δώσετε να απευθυνθώ στην Επιτροπή σα Να αναφερθώ επίση στο ότι είμαι και πρόεδρο ε, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και πέρσι δημοσιεύσαμε μια έκθεση πολιτικής για τη μεταρρύθμιση της ρύθμισης των αγορών με επικεφαλής τον Μάρτιν Χέλβιχ. Θα βρείτε και παραπομπή στην έκθεση αυτή, στις ε, σημειώσεις μου. Θα ήθελα να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση των ζητημάτων και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε για το ποιος είναι ο στόχος του νέου αυτού ρυθμιστικού πλαισίου που είναι, δηλαδή να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας συστημικής ε, κρίσης ε, που από ό,τι φαίνεται ακόμα συνεχίζεται με ένα κόστος που έχει υπολογιστεί ε, γύρω στο 8% του ΑΕΠ της Ένωσης τα έτη 2007 μέχρι 2010 χωρίς να συμπεριλάβουμε δηλαδή την τρέχουσα κρίση. Το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι πως από ό,τι φαίνεται ένα πολύ μικρό πρόβλημα στην αγορά των στεγαστικών των ΗΠΑ. δημιουργήσε μια τεράστια κρίση και το θέμα είναι το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και το επιχείρημα είναι πως οι υψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει μπορούν να περιορίσουν τους ε, κινδύνους συστημικών κρίσεων στο παρελθόν. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη πως δεν μιλάμε μόνο για την σταθερότητα μεμονωμένων ιδρυμάτων ε, στο σύνηθες ε, μακροπολιτικό πλαίσιο, αλλά μιλάμε για τη σταθερότητα του ίδιου του συστήματος και το πρόβλημα με το τωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο είχαμε μέχρι τώρα είναι πως ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα γιατί πάρα πολλές τράπεζες είχαν μειώσει το κεφάλαιό τους σε ένα ποστό 1 έως 3% των συνολικών τους ε, στοιχείων ε, ενεργητικού σταθμισμένα πάντα για τον ε, κίνδυνο. Οπότε, με κακοπρόθεσμα θα πρέπει να αποκαταστήσουν την κεφαλή επάρκεια και να πουλήσουν αρκετά στοιχεία τους και έτσι δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Εάν λοιπόν αυξήσουμε τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. το αποτέλεσμα αυτής της απομόχλευσης θα είναι πολύ μικρότερο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θα αυξήσουμε π.χ. το κεφάλαιο σε ένα 15% του συλλογισμού των τραπεζών, οπότε έχουμε... Ε, ένα ποσό των 6,7 ε, ευρώ ε, ευρώ το οποίο θα πρέπει να απολυθεί για να αποκαταστήσουμε ένα ευρώ ζημιά. Οπότε γι' αυτό ζητάμε υψηλότερε κεφαλιακές απαιτήσει και μάλιστα κατά την άποψή μου οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται δεν πηγαίνουν αρκετά μακριά όσον αφορά την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Είναι δύσκολο το να πούμε το ποια θα είναι η επαρκή κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα Βεβαίω μιλάω για μέσο μακροπρόθεσμε λύσει, γιατί πάρα πολλά για ε, επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη σε κρίση και τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Οπότε εγώ θα έλεγα πως θα πρέπει να πάμε ακόμη ψηλότερα από τον, την τωρινή αναλογία μόχλευσης και να εξετάσουμε ένα υψηλότερο ποστό του κεφαλαίου στο σύνολο του ισολογισμού χωρίς να είναι σταθμισμένο για τον κίνδυνο. Επίσης, όταν μιλάμε πως αυτή θα είναι η λύση για το πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού τομέα, δεν επαρκούν μόνο οι κεφαλαιακές απαιτήσει, είναι κοντόφθαλμο να λέμε κάτι τέτοιο. Χρειάζονται πολλές συμπληρωματικέ μεταρρυθμίσεις και όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα καθώς επίλυση το οποίο θα αντιμετωπίζει το ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια αναγκαστική επανακεφαλαιοποίηση ή να κινητοποιήσουμε τις τράπεζες για να αυξήσουν το επίπεδο κεφαλαιοποίησης ε, μέσω των αγορών. Και βεβαίως ο δεύτερος πυλώνας ε, του πλαισίου της ε, Βασιλείας είναι η δυνατότητα να, αυξηθεί, να αυξηθούν οι διακριτικές εξουσίες οι οποίε ε, υπάρχουν στι ρυθμιστικέ αρχέ. Κατόπιν δεν θεωρώ πω οι υψηλότερε κεφαλαϊκέ απαιτήσει κοστίζουν. Εγώ θα έλεγα πω μειώνουν τον κίνδυνο συστημικής κρίσης και βεβαίως το κόστος της συστημικής κρίσης είναι τεράστιο, οπότε αν βρεθεί ένας τρόπος να το μειώσουμε, νομίζω πως αυτό είναι υπέρ των υψηλότερων κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Επίσης λέμε συχνά πως τράπεζες με υψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει δανείζουν λιγότερο. Δεν το βλέπω. Βασικά μπορούμε να έχουμε διάφορες προσαρμογές στους λογισμούς. Εάν π.χ. αυτές οι απαιτήσει επιβληθούν σε βάθος χρόνου, όπως προγραμματίζεται, υπάρχουν επίσης εμπειρικά στοιχεία που μας δείχνουν πως ο αρνητικός αντίκτυπος στον τραπεζικό δανεισμό δεν είναι ε, ο αναμενόμενος. Επίσης, υπάρχουν πολλές εμπειρικές μελέτες για αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο να βρούμε στοιχεία που δείχνουν μεγάλη αύξηση στο κόστος ε, δανεισμού ή στο κόστος μετοχικού κεφαλαίου. Αλλά οπωσδήποτε μέσω μακροπρόθεσμα θα έχουμε μία μετατόπιση στην ε, δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε χρηματοδότηση περισσότερο μέσω μετοχικού κεφαλαίου. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά την στάθμιση κινδύνου των κρατικών ομολόγων με μηδέν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την αξιολόγηση κινδύνου και το πώς καλά είναι τα μοντέλα μας. Οπωσδήποτε δεν προσπαθώ να αξιολογήσω τον κίνδυνο που υπάρχει για τους συλλογισμούς των τραπεζών και έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει μια ακριβής ε, μέτρηση και αξιολόγηση. Το θέμα το οποίο βρίσκω εγώ προβληματικό είναι πως ε, το μοντέλο κινδύνου μίας τράπεζας εξορισμού δεν μπορεί να λάβει υπόψη τα συστημικά αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης ε, παραμέτρου απλούστατα γιατί μια τράπεζα δεν έχει αυτές τις πληροφορίες από μόνη της και όλοι γνωρίζουμε βεβαίως το ποιο είναι το πρόβλημα αν έχουμε κρίση σε μια τράπεζα συστημικής σημασία. Οπότε για την κατάσταση την οποία σκεφτόμαστε, δηλαδή ένα γεγονό συστημικού κινδύνου στις ε, χρηματαγορές, δεν νομίζω πως τα μοντέλα κινδύνου που έχουμε επαρκούν για να εξετάσουν αυτή την ε, κατάσταση. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για την δυνατότητά μας να μετρήσουμε τον κίνδυνο στους συλλογισμούς των τραπεζών. Νομίζω λοιπόν πως ε, είναι σχετικά σαφές πως η μηδενική στάθμιση κινδύνου για δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα που υπάρχει στις αγορές και νομίζω επίσης πως εάν σκεφτούμε και τα στοιχεία που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου, αν η τράπεζα αποφασίζει αν θα επενδύσει σε δημόσιο χρέος ή σε επιχειρηματικό χρέος, ο μηδενικός κίνδυνος είναι κίνητρο για να επενδύσει σε δημόσιο χρέος εντός μιας συγκεκριμένης κλάσης κινδύνου, οπότε θα πρέπει να φύγουμε από την μηδενική αξιολόγηση κινδύνου των ε, κρατικών ομολόγων. Να αναφέρω και κάτι άλλο, το τέταρτον, το τι είναι ο συστημικός ε, κίνδυνος και αν θεωρούμε πως σχετίζεται μόνο με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Βεβαίω, ναι, αυτό είναι το προφανέ. Μια τράπεζα που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα τη ή για, τον, ε, για το κομμάτι τη αγορά τη ε, και μόνο λόγω του μεγέθου τη έχει συστημική σημασία. Μπορεί όμω να είναι πιο συνδεδεμένη επίση με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από μια μικρότερη τράπεζα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πω και μικρέ τράπεζε μπορούν να έχουν συστημική σημασία. Αυτό ισχύει εάν είναι εκτεθειμένες όλες στους ίδιους μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνους. Εάν πολλές, πολλά μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι εκτεθειμένα στους ίδιους μακροοικονομικούς κινδύνους και αρχίζουν να υποφέρουν π.χ. αν αυξάνονται τα επιτόκια αναχρηματοδότησης, αυτό θα έχει επίσης συστημικό αποτέλεσμα. Και βλέπουμε παραδείγματος χάρη τι έγινε στην Αμερική με τις savings and loans, τα ιδρύματα αυτά, όπου δεν ήταν αρκετά μεγάλα για να, είναι σε, να θεωρηθούν σημαντικά για το σύστημα, παρόλα αυτά προκάλεσαν μια σημαντική κρίση. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητής είναι ο Τιέρη Φιλιππονά, Γενικός Γραμματής του Finance Watch. Καλό μεσημέρι. Τη Finance Watch θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή Οικονομικών και Νοσηματικών Θεμάτων ε, που μας κάλεσε να συμμετάσχουμε στην ακρόαση αυτή. Εν μέσω των τελευταίων χρηματοοικονομικών αναταράξεων, οι ηγέτες της Ευρώπης εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός σχεδίου αναχρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Νομίζουμε ότι είναι επίγουσα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίγουσα η ανάγκη οικοδόμησης ενός πιο ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος Η θέση του Finance Watch ό,τι αφορά τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει των τραπεζών θα μπορούσε να συνοψιστεί Ω εξή. Πρώτα απ' όλα, υψηλότερο κεφάλαιο τραπεζικό δεν βλάπτει την ικανότητα των τραπεζών να ε, προβούν σε δάνειο προς την πραγματική οικονομία. Δεύτερον, μια, ένας απλός λόγος θα πρέπει να είναι το βασικό ρυθμιστικό εργαλείο για το τραπεζικό κεφάλαιο. Και τρίτον, οι λόγοι που βασίζονται σε στάθμιση κινδύνου θα πρέπει να είναι ένα δευτερεύον εργαλείο για τη βελτίωση τη τραπεζική εποπτεία και θα επανέλθουμε. Το Finance Ghost θεωρεί επίση ότι σε ό,τι αφορά την αντοχή των τραπεζών, η ρευστότητα είναι εξίσου σημαντική με το κεφάλαιο. Το βασικό συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε από τι χρηματοοικονομικέ αναταράξει των προηγούμενων ετών είναι ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή ένα σύστημα που θα είναι και αποδοτικό και ανθεκτικό. Δύο ερωτήσει λοιπόν πρέπει να ε, θέσουμε. Η ΟΚΑ 4 θα κάνει πιο αποτελεσματικέ, πιο αποδοτικέ τι ευρωπαϊκέ τράπεζε, είναι το πρώτο ερώτημα. Ένα σημαντικό στοιχείο ε, τη αποδοτικότητα ε, έχει να κάνει με το κατά πόσο οι υψηλότερε κεφαλαϊκέ απαιτήσει θα αυξήσουν το κόστο χρηματοδότηση των τραπεζών και θα μειώσουν τη δυνατότητα ε, δανειοδότηση προ την πραγματική οικονομία. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα σύντομο όχι ότι δηλαδή η δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών δεν επηρεάζεται από το μείγμα χρέους ε, και χρηματοδότηση το οποίο θα επιλέξουν. Και ε, αυτά τα αποδεικνύει και η θεωρία και, η εμπειρική, ε, και τα εμπειρικά στοιχεία. Μπορώ όμως να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας στη συνέχεια. Εάν τώρα πρέπει να υπάρξει απομόχλευση από τι τράπεζε ώστε να συμμορφωθούν προ το ΟΚΑ 4, δεν θα πρέπει να μειώσουν τα δάνεια προ την πραγματική οικονομία. Μπορούν να απολύσουν άλλα στοιχεία ενεργητικού, όπως το χάρη παράγωγα ή χαρτοφυλάκια ε, trading, συναλλαγών, που είναι κατά μέσο όρο το δύο, τα δύο τρίτα του ισολογισμού των μεγάλων ε, ευρωπαϊκών τραπεζών. Δεύτερο ερώτημα σε σχέση με την αποδοτικότητα είναι κατά πόσον ε, ο ΟΚΑ 4 θα δώσει δυνατότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες ε, να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς μεταξύ του πελάτες. Ένα αποτελεσματικό, ένα αποδοτικό τραπεζικό σύστημα δίνει στις τράπεζες την ελευθερία να αποφασίσουν ποια στοιχεία ενεργητικού θα χρηματοδοτήσουν. Αν χρησιμοποιηθεί ως βασικό ε, πρωταρχικό ρυθμιστικό εργαλείο η στάθμιση κινδύνου, όπως γίνεται με την ΟΚΑ 4, ε, τότε όλες οι τράπεζες αναγκάζονται ουσιαστικά να έχουν τα ίδια στοιχεία ενεργητικού ε, στην κατοχή τους. Και δίνει την εντύπωση, που είναι αυταπάτη όμως, ότι μπορεί η αξιολόγηση κινδύνου ουσιαστικά να ε, οριστεί μόνο με ένα νομοθέτημα και κάποια α, στοιχεία ενεργητικού, πάντοτε είναι πιο επικίνδυνο. Γίνεται και λιγότερο διαφοροποιημένο και λιγότερο αποδοτικό το σύστημα. Τώρα, ποιο ε, θα ήταν το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών ε, με την ΟΚΑ 4. Τρία, υπό τρία διαφορετικά πρίσματα μπορούμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, εάν θα μπορέσει η ΟΚΑ 4 να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές τράπεζες αυτόνομες. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί. Όπως προϋπόθηκε, η ποιότητα των κύριων δύο κεφαλαίων, το Equity Tier 1 Capital, βελτιώνεται σε ό,τι αφορά την ΟΚΑ 4, ε, σε ό,τι αφορά ιδίω ε, την ε, ικανότητα απορρόφησης απολειών. Το ποσοστό κεφαλαίου που απαιτείται από τις τράπεζες από το 2% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού πηγαίνει στο 4,5% και ίσως φτάσει και στο 7%. Εδώ, σε ό,τι αφορά τώρα τις απαιτήσει ρευστότητα, ε, θα είναι, πιο, θα είναι λιγότερο έφταυστε οι τράπεζες ε, χάρη στην ΟΚΑ4. Το είδαμε με τη Lehman Brothers, την Northern Rock, τη Ford, τη Dexia Bank, πόσο σημαντική είναι η ρευστότητα. Το ίδιο σημαντική με, το, με την επάρκεια κεφαλαίου των τραπεζών. Και νομίζουμε ότι είναι οικονομικά λογικός ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι παρονομαστές ε, των λόγων ε, ρευστότητας. Και επίσης ό,τι αφορά την ε, απλή, τον απλό λόγο μόχλευσης, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι πρωταρχικό εργαλείο και θα επανέλθουμε. Είναι απλό πάντως και αποτελεσματικό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Θα μπορούσε να πάει τόσο μακριά όσο Θέλουμε στο, στην δημιουργία ανθεκτικών τραπεζών το ΙΟΚΑ4. Απαντάμε όχι σε αυτό το ερώτημα. Πρώτον, γιατί ναι, μεν έχουμε αυτή την αύξηση των βασικών ιδιών κεφαλαίων από το 2 στο 4,5%, αλλά αυτό ουσιαστικά ισοδυναμεί με το 2% του συνολικού ισολογισμού. Και θα πρέπει να συγκριθεί αυτό με τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται για τη Lehman Brothers, παραδείγματο χάρη, η οποία πρωτού πτωχεύσει είχε 11% αναλογία βασικών ίδιων κεφαλαίων. Και για την τέξια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 10,4% τον Ιούλιο του 2011. Άρα πηγαίνουμε ε, όσο μακριά πρέπει, όχι. Νομίζω ότι απαντάει στο ερώτημα ε, το παράδειγμα το οποίο σας ανέφερα. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τον, ε, την αρχή οποία, στην οποία βασίζεται η Βασιλεία Τρία, δηλαδή το value at risk, είναι μια μέθοδος που έχει κάποια πλέον αλλά δεν ωφελεί σε περίοδο κρίσης να χρησιμοποιούμε αυτό το γνώμονα. Η μέθοδος δηλαδή πολιτισμό που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να αποδώσει εν καιρό κρίσης. Τρίτος λόγος για τον οποίο απαντάμε όχι είναι ότι οι σταθμίσεις κινδύνου σε μεγάλο βαθμό αποτελούν ε, την απόρρεια εσωτερικών τραπεζικών υπολογισμών. Άρα μπορεί τα ίδια στοιχεία κινδύνου να δώσουν τελείως διαφορετικές σταθμίσεις κινδύνου ανάλογα με την τράπεζα. Άρα ουσιαστικά δεν έχει νόημα αυτό το headline capital ratio για τους επενδυτές και τους ρυθμιστές. Άλλο ερώτημα, θα συμβάλλει ο K4 στην οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος, γιατί πριν είδαμε τις μεμονωμένες τράπεζες κατά πόσο μπορεί να γίνουν πιο ανθεκτικές. Τώρα κοιτάμε το όλο σύστημα. Και ίσως είναι και το σημαντικότερο ερώτημα αυτό, τελευταίο. Με την χρησιμοποίηση σταθμίσεων κινδύνου ως πρωταρχικό ρυθμιστικό εργαλείο, η ΟΚΑ 4 όχι μόνο δεν βελτιώνει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά την δυσυραίνει, την επιδεινώνει. Και ποιο είναι ο λόγο γι' αυτό. Οι σταθμίσει κινδύνου ουσιαστικά είναι ένα κίνητρο για τι τράπεζε να αυξήσουν την αλληλοσύνδεσή του. Και ένα πιο αλληλένδετο εξορισμού σύστημα είναι και πιο εύθραυστο. Πώς λειτουργεί όλο αυτό όταν μια τράπεζα αγοράζει, αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο ή κάνει ένα ε, δάνειο. Μπορεί να μειώσει το ποσό του κεφαλού που πρέπει να έχει χρησιμοποιώντας ε, παράγωγα. Παράδειγμα η IAG. Στην ετήσια έκθεση του 2007 έγραψε η εταιρεία ότι 379 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου ε, ασφαλίστρων κινδύνου είχαν πολιθεί σε χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Θα διαβάζω μέσα από την έκθεση. Κυρίω στην Ευρώπη. Και ο στόχος δεν ήταν τόσο ο μετριασμός του κινδύνου, αλλά κάποια ανακούφιση ότι αφορά το ρυθμιστικό, ρυθμιστική, ανακούφιση, ρυθμιστική κεφαλαϊκή ανακούφιση. 379 δί Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το αρμπιτράζ να αλλάξει με, το, με τη Βασιλεία 3 ή με το ΟΚΑ 4. Έρχομαι σε κάποια συμπεράσματα. Για να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που θα χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητα και ανθεκτικότητας χρειαζόμαστε governance, διακυβέρνηση. Ποια είναι τα βασικά μας μηνύματα. Πρώτον, δεν βλάπτει την πραγματική οικονομία το μεγαλύτερο τραπεζικό, η αύξηση του τραπεζικού κεφαλαίου. Δεύτερον, απλώς, απλώς λόγος μόχλευσης, αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο για να πετύχει ο διτός στόχος αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας. Και τρίτον, για να μην έχουν περιβολική συσσόρευση κινδύνου Μόνο υποστηρικτικό ρόλο πρέπει να έχουν οι σταθμίσει κινδύνου. Η χρήση λοιπόν ε, σταθμίσεων κινδύνου, όπω είδαμε, ω πρωταρχικού μηχανισμού δεν είναι αποδοτικό και επίση αυξάνει και το συστημικό κίνδυνο, τη συνολική μόχλευση και την ομοιογένεια των στοιχείων του ενεργητικού. Μία βασισμένη στον κίνδυνο ε, προσέγγιση είναι κατάλληλη ταυτόχρονα για του επόπτε για να κατανοηθούν οι κίνδυνοι και να μπορούν αυτοί να παρεμβαίνουν ε, όπου δει. Μία τώρα αμυγής προσέγγιση μόχλευσης θα μπορούσε να έχει ω αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου στι τράπεζε εντό των περιορισμών μόχλευση. Το είδαμε και με τη Βασιλεία 1. Άρα θέλουμε συνδυασμό τη αμυγού μόχλευση και των σταθμίσεων κινδύνου. Αλλά καλό θα ήταν η σχέση μεταξύ μόχλευση και σταθμίσεων κινδύνου να ε, αντιστραφεί. Δηλαδή πρωταρχικό κανόνα να είναι η μόχλευση. Τέλος, ό,τι αφορά το λόγο αυτόν, ε, το, 30, το επί 33, το λόγο μόχλευσης που αναφέρεται στο K4, ε, ουσιαστικά χάνεται οποιοδήποτε οικονομικό στόχος, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό. Εμείς θα κάνουμε προτάσεις να είναι πιο λογικό οικονομικά το όριο αυτό και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι ε, και ο ιστικός κίνδυνο ε, και το λεγόμενο too big to fail για τις τράπεζε, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να μην καταρρεύσουν και άλλε τράπεζε. Ευχαριστώ τελευταίο ομιλητής Richard Reburn, πρόεδρο του European Association of Corporate Treasurers. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην δημόσια ακρόαση. Είναι ζωτική σημασία οι σχέση της πραγματική οικονομίας ε, και του συστήματος να εισακούγονται οι απόψει από του νομοθέτες. Έχουμε ενώσει τραπεζικές από 17 κράτη-μέλη που συνέρχονται σε αυτό το πλαίσιο και την Ελβετία και την Κροατία. Είμαστε επαγγελματίε, δεν είμαστε ενώσει ε, εμπορίου και δεν ασκούμε λόμπι τομεακά, δεν έχουμε κανένα κέρδος ε, για κάποια εμπορική προώθηση συμφερόντων. Ενδιαφέρον μας είναι η επαγγελματική προαγωγή της, ε, του πλαισίου όσον αφορά τον δανεισμό και τις ε, λειτουργίες μας. Βρήκαμε όλο και περισσότερο ότι ανθρώνουμε την φωνή μας ε, για την πραγματική οικονομία. Το να αναγνωριστεί η φωνή αυτή είναι μια ανάγκη που είναι πραγματικά επιτακτική για τον τομέα αυτόν και για τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν. Αυτές οι παρουσιάσεις ε, ξεκινούν πάντα με μια επιβεβαίωση για το έργο των νομοθετών να σταθεροποιήσουν ε, το σύστημα σωστά εστιαζόμαστε στο να προστατευτούν οι σημερινές και μελλοντικές γενναίες ε, από τις αρνητικές επιπτώσεις όσων πάνε στραβά και μπορούν να αποτύχουν. Όμως ο εστιασμός πρέπει να βρίσκεται στα πραγματικά αίτια της κρίσης, ενώ η κακή νομοθεσία προφανώς δεν βοηθά καθόλου οι ρυθμίσεις που δεν ταυτοποιούν τα πραγματικά αίτια και που πραγματικά αγνοούν τον εντοπισμό των αιτίων της ε, κρίσης ε, βλάπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ολόκληρη σειρά επιπτώσεων. Αυτές οι επιπτώσεις ε, είναι εκείνες που μας οδήγησαν να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά τα παράγωγα, για παράδειγμα, και τι ρυθμίσει άλλαξαν σημαντικά οι αρχικές ε, προτάσεις όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Χαιρόμαστε για την ε, συμπερίληψη αυτών των ρυθμίσεων και των εξαιρέσεων. Επικεντρώνουμε στις παρατηρήσεις μας σε κάποιες πτυχές της πρότασης για το CRD4 την ε, οδηγία για κεφαλαιακή επάρκεια δηλαδή και τι επιπτώσεις ε, στην πραγματική οικονομία, τι μεγάλες ε, εταιρείε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, η συνεκτικότητα και συνάφεια όσον αφορά την ΟΚΑ 4 από πλευρά του 2009 και του Σεπτεμβρίου για τι συμβάσει και ενιοποιημένα πλαίσια την υποβολή εκθέσεων υποχρεωτικά και την αποσαφήνιση οποια, οποιονδήποτε εκκρεμούντων παραγωγών. Όταν ξεκινήσαμε, σωστά τονίστηκαν οι σοβαρές, ε, χωρίς πρόθεση όμως αρνητικές επιπτώσεις. Στην μεταρρύθμιση του, της Βασιλείας 3 που συνέχισε το αρχικό έργο, Υπάρχουμε, υπάρχει εκεί και μια αντίφαση όσον αφορά την τελική έκβαση. Συγκεκριμένα, αν προχωρήσει το CRD4 όπως ε, έχει σχεδιαστεί, οι επιπτώσεις ε, στα παράγωγα θα μπορούσε να είναι αρνητική και να είχαμε ε, το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλησαν οι νομοθέτες και είχαν συμφωνήσει και εδώ αλλά και στην Ουάσιγκτον. Στις συζητήσεις αυτές προσπαθήσαμε να τονίσουμε ότι ο συστημικός κίνδυνος ε, δεν προέρχεται, ε, ε, συναρτάται με την ελλειπή αντιμετώπιση των αιτίων. Και θα πρέπει εδώ να δούμε και το κατά πόσον αυτή η αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου μπορεί να ενταχθεί στις προτάσεις. Μεγαλύτερη κεφαλιακή επάρκεια μπορεί να προστατεύσει από αυτούς τους κινδύνους χωρίς όμως συνάρτηση μεταξύ συστημικού κινδύνου και αναχέτησης του κινδύνου από συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όσον αφορά τις συναλλαγές και τις συναλλαγές με παράγωγα. Γι' αυτό το CRD4 για την τιμή των παραγώγων όσον αφορά τους υπολογισμούς είναι ένας πάρα πολύ τεχνικός τομέας και θα ήθελα τρία σημεία να τονίσω εδώ. Η προηγμένη ε, προσέγγιση που ε, λαμβάνει υπόψη τα CDS και την βάση υπολογισμού και την περίοδο ε, κάλυψης ε, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παραγωγά. Μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση από ότι το, το αντίστοιχο ε, χωρίς το CDS θα κόστιζε. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη δεύτερον. Η συμπερίληψη των στοιχείων CDS στους υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανησυχίες που υπάρχουν είναι σημαντικό στοιχείο και από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου ο υπολογισμός συμπεριλαμβάνει στοιχεία και διπλής ε, λογιστικής. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία ε, περιέγραψα δεν θα, είχε, δεν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις ε, αν ήταν μόνο θεωρητικά, στο θεωρητικό επίπεδο και όχι στην πραγματική οικονομία. Σε αυτή τη φάση εκτιμήσεις όσον αφορά τις τιμές επιβάρυνσης των παραγωγών κυμαίνονται. Όμως η επιβάρυνση θα μπορούσε να διπλασιάζεται όσον αφορά το αρχικό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για την πραγματική οικονομία και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να γίνει η προσπάθεια αναχέτησης, μείωση αυτού του κινδύνου. Οδηγούμαστε στη δεύτερη πτυχή του CDR4 και τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Όσον αφορά τις αντικές επιπτώσεις για το κόστος, για τις επιπτώσεις που θα υπήρχαν στο κόστος και για την χρήση των παραγόγων υπάρχουν και άλλοι τομείς ανησυχίας. Σύντομα θα καλύψω τους εξής τομείς. Αυτό που θα κάνει το CDR4 στο κόστος δανεισμού θα ασκηθεί πίεση στις μικρότερες ε, ε, εταιρείες που δεν έχουν και δεν θα έχουν πρόσβαση στις κεφαλαϊκές αγορές. Και έχουμε και θέματα διεθνούς ανταγωνισμού που αναφύονται οι επιπτώσει στο κόστος δανεισμού είναι δύσκολο να ποσοστοποιηθούν. Μια ομάδα γερμανικών ε, επιχειρήσεων ζήτησαν να υπάρξει μια μελέτη που θα συνταχθεί για αυτά τα στοιχεία. Είναι πρόδειλο, παρότι έχουν ακουστεί διάφορα επιχειρήματα, ότι το κόστος θα αυξηθεί. Η Standard Poor's δημοσίευσε μια μελέτη με βάση την Βασιλεία 3 μεταξύ 50 και 60 μονάδων βάσης ε, σε σχέση με την επιβάρυνση ανάλογα με την φερεγγιότητα του ε, ε, δανειζόμενου και την σχέση του με τα τραπεζικά ιδρύματα. Χωρίς αυτή την αναλογία το βάρος του πρόσθετου δανεισμού θα είναι από 20 μέχρι 142 μονάδες βάσης για εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται από τον τραπεζικό δανεισμό Αυτές είναι σημαντικές επιβαρύνσεις. Θα αυξήσουν το συνολικό κόστος κεφαλαίου συνολικά και θα καταστήσουν τις ε, ε, σωστές ε, αποτελεσματικές επενδύσεις δυσχερέστερες. Θα έχουμε αύξηση στο άκρο του φάσματος που μόλις περιέγραψα και θα αλλάξει η ε, χρηματοδότηση όσον αφορά τις ε, τράπεζες, μεγάλες τράπεζες και την αγορά. Αυτό δεν είναι επικοδομητικό σε περίοδο ανάκαμψης, οικονομικής ανάκαμψης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται ιδιαίτερα από την προοπτική αυτή απομόχλευσης, ε, απομοχλικής δράσης όσον αφορά τις τράπεζες στη χρηματοδότηση του εμπορίου, των εμπορικών δράσεων, είναι ενθαρρυντικό ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστούν πιο υποφελείς προοπτικές ε, ε, όσον αφορά την αναθεώρηση του πλαισίου της Βασιλείας 3. Έχουμε θέματα ε, ρευστότητας, ε, μοχλικής επίπτωσης ε, σε σχέση με την ε, Βασιλεία 3 και την αναθεώρηση με βάση τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Οι οικονομικές αυτές προοπτικές φαίνεται ότι υπερβάλλουν όσον αφορά τον κίνδυνο της χρηματοδότησης των εμπορικών αυτών συναλλαγών και την έκθεση τραπεζικών, τραπεζών σε κινδύνους. Θα πρέπει εδώ να δούμε και τις πιστώσεις στα δάνεια για τις εξαγωγές. Όπως προτείνεται, οι εγγυήσει δεν προβλέπουν κάποια αλλαγή όσον αφορά την κεφαλαϊκή επάρκεια. Αυτός ο τομέας θα καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εποπτείας Τραπεζών Ελπίζουμε ότι το καθεστώς CDA4 δεν θα καθοριστεί τελεσίδικα προτού υπάρξει υποβολή έκθεση σχετικά. Το θέμα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας αναφύεται όσον αφορά ένα ισοδίκαιο πλαίσιο και πεδίο δραστηριοποίησης και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πτυχές που προανέφερα και μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις εξαγωγές και τις πιστώσεις προς τις εξαγωγές. Αν δεν ληφθούν αυτά υπόψη θα αποβούν εις βάρος των εξαγωγέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, πρέπει να δούμε ότι πολύ περισσότερο έχουν παγιωμένη θέση ε, η ΕΠΑ Πράγμα το οποίο αν υιοθετηθεί γενικά αυτή η προσέγγιση της Βασιλείας 3 θα είναι προς όφελος αυτών των ε, εταιριών. Έχουμε και ένα νέο κεφαλαιακό καθεστώς για μια νέα χρηματοοικονομική σταθερότητα, σταθεροποίηση και αποτελεσματικότητα τραπεζών που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Αυτό μπορεί να υποφελήσει εταιρείε που υποφελούνται από νέε αγορέ. Ωστόσο δεν θα είναι προ όφελο όλων. Οι ανησυχίε που εκφράζονται για το CAD4 και τη Βασιλεία 3 είναι ανησυχίες και μελήματα που συμμερίζονται ευρέως η μετοχή μα και οι εμπλεκόμενοι στον τομέα. Έχει απευθυνθεί και επιστολή από πολλέ εταιρείε που εφιστά την προσοχή στι μη θελημένε επιπτώσει όσον αφορά τα παράγωγα για παράδειγμα η ACT έχει πάρα πολλές εταιρείες ε, που δεσμεύονται να προσθέσουν ε, τις, ε, τα ονόματά τους, την επωνυμία τους σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ελπίδα μου ότι η ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την ακρόασή σας και η επιστολή μας θα συνεισφέρουν να είναι υποφελής η έκβαση αυτών των προσπαθειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προσβλέπω στο να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Πρέπει να πω πως άκουσα πάρα πολλά πράγματα που συμφωνούν με αυτά τα οποία λέω και να κάνω σκέφτομαι πως πρέπει να προχωρήσουμε με την νομοθεσία για την τέταρτη οδηγία εκφυλακών απαιτήσεων. Η Βασιλεία 3 ακόμα είναι υπό επεξεργασία. Το ξέρουμε πως θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε ορισμένους τομείς και ίσως υπάρχουν κάποιοι τομείς ο θα πρέπει να γίνει αυτό τώρα για τους ομιλητές. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Ζαν Πολ Κλίντς, Γκίγκολτ, Βίκυ Ότμαρ, προφανώς. Ποιος άλλος? Ο Πασκάλ. Ο ένας αντί για τον άλλον, τι θέλετε. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Εγώ δεν θα παρέμβω. Έχουμε πάνω από μία ώρα. Εάν θέλετε βεβαίως να απαντήσουν όλοι σε όλες οι ερωτήσεις θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Οπότε τι θα κάνω. Θα ακούσουμε πολλές ερωτήσεις και μετά θα ζητήσω από το πάνελ ε, να σημειώνει βεβαίως ε, το πώς θα απαντήσει. Αναρωτιέμαι. Ότμαρ, θέλετε εσείς πρώτος όσοι είστε να μιλήσετε ή θέλετε να ακούσετε πρώτα τους υπόλοιπους. Ωραία. Ο, με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο. Οπότε ο Ζαν Πολ έχει πρώτος ο λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές οι οποίοι διαφώτισαν με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το θέμα αυτό και προσπάθησαν να είναι σαφείς στις παρεμβάσεις τους. Κάτι το οποίο αποτελεί ποιότητα για το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, την πρώτη επίσημη ε, παρουσίαση του, Finance, ε, του Financial Watch, στρέφομαι στον εκπρόσωπο του. Θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχουν αντίβαρα στο επίπεδο του lobbying και με υπέρ του lobbying προσωπικά και να υπάρχει κάποια ισορροπία. Θέλω λοιπόν στον κύριο Φιλιππονά από το Finance Watch να θέσω το εξή ερώτημα. Αν σα κατάλαβα καλά, είπατε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα αυστηρό περιορισμό, ένα αυστηρό όριο στη μόχλευση. Το ερώτημά μου το εξή. Ένα τέτοιο όριο, μήπω ε, θα αποτελούσε έναν αρνητικό κίνδυνο επί τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Επειδή ήταν πολύ απλό, γλυκό και αποτελούσε ερώτημα προς έναν μόνο από εσάς, σας δίνω το λόγο να απαντήσετε. Κύριε Κοζέ, σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι να απαντήσω ε, θα πρέπει και μπορούμε ήδη να το βάλουμε αυτό το ερώτημα σε προοπτική. Αν δούμε τους λογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών, των μεγαλύτερων τραπεζών, εκεί βλέπουμε, ε, καλά για τις μικρότερες έχουμε ένα πραγματικό θέμα, αλλά όταν βλέπουμε τον ισολογισμό των μεγαλύτερων ε, τραπεζών, τα δύο τρίτα του ισολογισμού δεν αντιστοιχούν σε δάνεια προς την πραγματική οικονομία. 70% είναι trading παράγωγα και 30% αντιστοιχεί στο, στα δάνεια, στα loans. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούμε απόλυτα λογικά να φανταστούμε αυτό τη μόχλευση ότι μπορούμε να μειώσουμε το πορτοφόλιο trading και παραγόγων, να πρόκειται για δραστηριότητε άλλωστε που δεν συμβάλλουν ή συμβάλλουν πολύ λίγο στη χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία και να κρατήσουμε τα δάνεια προ τι επιχειρήσει. Γνωρίζω βέβαια ότι το επόμενο ερώτημα είναι ναι, αλλά αν έχω ένα καλύτερο return on equity, καλύτερη απόδοση κεφαλαίου, μπορώ να μειώσω ε, τα δάνεια στην πραγματική οικονομία, διότι βελτιώνω ό,τι έχει να κάνει με τα ίδια κεφάλαια στο Book of Trading. Αλλά ε, ένα παράδειγμα, η απόδοση κεφαλαίου ε, για τη δραστηριότητα Delta 1, Delta 1 για την οποία μιλήσαμε με τη UBS, στο πλαίσιο της UPS. Όταν έχουμε το 50% απόδοση κεφαλαίου, επιστροφή φυσικά δεν είναι εύκολο. Αλλά αν δούμε το δημόσιο συμφέρον, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον ίσως να παρέμβουν οι ρυθμιστικές αρχές και να πούν στις τράπεζες ότι καλό το ΔΕΛΤΑ 1, υπάρχει καλή απόδοση κεφαλαίου σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια, αλλά θέλω να κάνετε μία ε, μείωση. Είδαμε τα προβλήματα πρόσφατα με μια λιβετική ε, τράψη και όχι να μειώσετε τα δάνεια στην πραγματική οικονομία. Είναι θέμα επιλογή. Αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχει όγκο. Υπάρχει όγκο για να μειώσουμε κάτι άλλο και όχι τα δάνεια στην την πραγματική οικονομία. Και αν είμαστε σε ένα σύστημα όπου ο μόνος νόμος ε, είναι απόδοση κεφαλαίου σε οικουμενικές τράπεζες που κάνουν και trading ε, και δανεισμό, για να τα πω απλά, πράγματι θα τεθεί το ζήτημα κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε σε αυτές τις τράπεζες κάτω από την ίδια στέγη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. I have a suspicion that the answer raises some... πως η απάντηση βεβαίω θα θέσει και άλλα ερωτήματα. Αν θέλει κανείς να επανέλθει, μπορεί αργότερα. Βολφ, κατόπιν. Ένα ερώτημα. να είναι επικριτικός για το ότι κάποιες τράπεζες όπως στην Ελβετία θέλουν να πάνε πολύ παραπέρα με τις κεφαλαιακές απαιτήσει από ό,τι προβλέπεται από τη φερικαιότητα. 4. Κανονικά διαμαρτυρόμαστε για τον ελάχιστο, όταν υπάρχει ο ελάχιστος κοινός ε, παρανομαστής. Τώρα από κάποιοι ζητάνε ψηλότερε απαιτήσει, γιατί διαμαρτυρόμαστε επίσης. Μην ξεχνάμε πως θα έχουμε και στον τομέα των ασφαλιών τη φερικαιότητα 2 και άρα θα πρέπει να δούμε και τη σχέση ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών και θα με ενδιαφέρει να ακούσω πώς το βλέπετε εσεί. Γιατί κάνουμε λάθο αν παριστάνουμε πώ δεν έχουν σχέση μεταξύ του οι δύο. Ε, I'm a little... Who is that? Αυτό σε ποιον απευθυνθήκε ακριβώς. Η, η τελευταία ερώτηση στην, ε, στην καθηγήτρια ή άλλη σε οποιονδήποτε. Okay, well, let's collect... Μάλιστα, ας ακούσουμε και την ερώτηση του Πασκάλ πρώτα για τους πράσινους. Εγώ είχα ένα ερώτημα προς ε, την κυρία Μπούχο, τον κύριο Φιλιππονά. Το πρώτο λιθαράκι της αξιολόγησης ε, κινδύνων που μετά σταθμίζεται είναι το κατά πόσο είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε με όσο τον πιο ακριβή τρόπο τους κινδύνους. Και οι κινδύνοι, τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες από όλους ε, τους σωματοπιστωτικούς ε, φορείς, λοιπόν, χρησιμοποιούν την νόμη των πιθανοτήτων. Κανονική νόμη αλλά τελείω διαφορετικά λειτουργεί η χρηματοπιστωτική αγορά. Από την Goldman Sachs, παραδείγματο χάρη, ο χρηματοοικονομικός διευθυντής λέει ότι το 2008 είδε πράγματα που με βάση του νόμου των πιθανότητων που χρησιμοποιούν τα μοντέλα, ε, στα μοντέλα του όλε οι τράπεζε, δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Όχι ότι θα ήταν λιγότερε πιθανότητε, ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορέ μεγάλε μεταξύ των κανονικών νόμων 25 αποστάσεις τύπου. Αν έχουμε μία μέρα ένα ε, συμβάν σε όλη τη ε, διάρκεια ε, ζωής του σύμπατος, έχουμε 8 διαστήματα τύπου. Εδώ μιλάμε για πολύ περισσότερα, δηλαδή αδύνατο να υπάρξει κάτι τέτοιο. μπορούμε να επεξεργαστούμε τα περιθώρια, τα... Ε, αλλά τι κάνετε στην περίπτωση αυτή. Αυτό το βασικό, το πρώτο λιθαράκι. Πώς μπορούμε να το καταστήσουμε χρήσιμο και ε, πώς μπορεί να βοηθήσει το ρυθμιστή και τον επόπτη να αξιολογήσει τον κίνδυνο. I think we've got time for people to come back on Νομίζω πως υπάρχει χρόνος. να επανέλθουν ε, οι αγορές. Πάντα θεωρούσα ότι οι οικονομικές αγορές ε, με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται υπάρχει το tunneling, το αποτέλεσμα προτού το αναμείνει κανείς ε, μπορεί να είναι δεδομένο. Αναμένουμε κάποιος να συντάξει μια διδακτορική διατριβή από αυτού. Τώρα έχουμε τις απαντήσεις ε, στις διάφορες ερωτήσεις ε, και ε, όσον αφορά τον Πασκάρ, Εσείς παρακαλώ. Για την πρώτη ερώτηση, για το ερώτημα γιατί δεν είναι καλό όταν τα κεφάλαια δεν αυξάνονται όπως και στις ελβετικές τράπεζες. Νομίζω το ίδιο θέμα είναι αυτό, όπως και για ένα περιορισμό ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο. Όσο υψηλότερο είναι, ο υψηλότερος είναι ο περιορισμός, τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Αν όλα τα αυτοκίνητα μόνο 20 χιλιόμετρα επιτρέπεται να τρέχουν, είναι λιγότερο επικίνδυνη οδήγηση. Όμως αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα αφέ αυτού. Και όπως ε, τονίστηκε, η, πως, η αναλογία ε, και πρόκειται μόνο για την ποσόστοση ως αναλογία αφορά μόνο τα αποθεματικά ή τα, το, κεφάλαιο των τραπεζών εν μέρη. Αυτό είναι που ασκούμε επικρίσεις ε, επ' αυτού. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι πέρα από αυτά την αξιολόγηση των, του ενεργητικού στους ισολογισμούς υπάρχουν ή μπορούν να υπάρχουν πολυάριθμα άλλα στοιχεία ενεργού κεφαλαίου που εξορισμού δεν έχουν κίνδυνο, όμως που γνωρίζουμε ότι τεράστιοι κίνδυνοι μπορούν να εμπεριέχονται. Και η UBS μπορεί να έχει 20% ε, ratio, αναλογία, αλλά σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνων ενεργητικού έχει πάνω από το δεκαπλάσιο όσον αφορά ε, περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους που όμως δεν έχουν αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο και έτσι δεν ε, μπορούμε να ε, το αποφύγουμε αυτό. Και γι' αυτό σε διαφοροποίηση με την άποψη πολλών συναδέλφων για την εισαγωγή μιας ευφυούς δράσεις εναντί της μοχλικής ε, ε, δράσης. Διότι αν μάθαμε κάτι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ή πρέπει να το έχουμε μάθει και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ε, τράπεζες αλλά και για τις ρυθμιστικές αρχές. Επιτρέπεται και οι ρυθμιστές να μαθαίνουν κάτι. Επιτρέπεται και οι ρυθμιστές να γίνονται σοφότεροι καθώς περνάει ο χρόνος. Ε, τότε θα πρέπει να έχουμε αναγνωρίσει ότι στους ισολογισμούς των τραπεζών υπάρχουν άπειροι, απειράριθμοι κίνδυνοι, ασύλληπτοι κίνδυνοι που μέσω της ποσόστοσης ή της αναλογίας δεν καλύπτονται. Και αυτό με οδηγεί στην προηγούμενη μου παρατήρηση, στο προηγούμενο σημείο μου. Τα ομόλογα της Ιταλίας έχουν μηδέν εκτίμηση κινδύνου. Αν όμως κανείς εκτός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αγοράζει τέτοια ομόλογα, ιταλικά ομόλογα, τότε έχουμε πραγματικά σοβαρότατο πρόβλημα. Εσείς νομίζω θα έπρεπε και εσείς να παρέμβετε. Yes, thank you very much. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Μόνο δύο λόγια έχω να πω για την ρευστότητα, την φερεγγιότητα η έκθεση που προανέφερα ότι συντάξαμε ουσιαστικά και μια σύντομη μελέτη που συντάξαμε για το Υπουργείο κάναμε λόγο για την Solvency 2 υπό την έννοια ότι στον μηχανισμό που έχουμε για τις ε, τραπεζικές ε, διατάξεις ε, και ε, κανονισμούς και το σύστημα πλαισίου. Ένα παρόμοιο μηχανισμό έχουμε στο Solvency 2. Οποτεδήποτε σκεφτόμαστε να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα κυκλικής επίπτωσης στον τραπεζικό τομέα, Πρέπει να δούμε υπό το Solvency 2 και υπό την, τις ρυθμίσεις για τις ασφαλίσεις ε, τι μπορεί να προκληθεί, τι μπορεί να γίνει. Και τα δύο ταυτόχρονα πρέπει να εξετάζουν και να καλύπτονται. Φυσικά οι ασφαλιστικές εταιρείε και οι τράπεζες κάνουν διαφορετικά πράγματα, αλλά εκ παραλλήλου πρέπει να βαίνει η αντιμετώπιση, η κάλυψη των κινδύνων. Τώρα και σε σχέση με την παρακολούθηση, εποπτεία κινδύνων, δεν λέω, γιατί έτσι ακούστηκε, σαν να λέγατε ότι η, ε, για την εποπτεία τραπεζών ότι ε, λέγαμε ότι κάτι είναι καλό ή μπορεί να μην είναι καλό. Εμείς λέγαμε ότι είναι θετικά όλα αυτά για τον στόχο για τον οποίο στοχεύουν να επιτύχουν. Δηλαδή την ε, δημιουργία ενός προφίλ κινδύνου για τις δραστηριότητες κάποιας τράπεζας ο λόγος για την ύπαρξη αυτών για μια τράπεζα είναι ένα κίνητρο να γνωρίζουν ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Αυτό όμως που έλεγα είναι κάπως διαφοροποιημένο. Ένα από αυτό είναι το ότι αναφέρθηκε ότι η περίοδος κρίσης ή η κατάσταση κρίσης είναι κάτι πολύ σπάνιο ως γεγονός και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες δεν έχουν στοιχεία για παρόμοιες περιπτώσεις κρίσης. Με βοήθεια λοιπόν για μια τέτοια πρόβλεψη πρέπει να συνεισφέρουμε να μπορούμε μπορέσουμε να έχουμε επαρκή στοιχεία για την πρόβλεψη αυτή ή την ε, ε, προοπτική αυτή. Και από την τράπεζα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, την τράπεζα της Αγγλίας, είναι ένα πρότυπο που συναρτάται από πάρα πολλές συνιστώσεις ε, σε σχέση με την ε, αναλογία κεφαλαίου που απαιτείται για την κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να καλυφθούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι. Μετά υπάρχουν διαφορές και διαφοροποιήσεις ε, όσον αφορά την δραστηριότητα των τραπεζών και αυτό δεν λαμβάνεται πάντα επαρκώς υπόψη. Και το τρίτο, και αυτό είναι και αυτό σημαντικό, η συνάρτηση μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε και από τα στοιχεία ΕΜΠΑ, ότι τα τραπεζικά συστήματα και οι διάφορες τράπεζες είναι σε υψηλό βαθμό συναρτημένες η μία με την άλλη, αλληλοσυνδέονται και σε περίπτωση που ε, δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία εργαζόμαστε με μάκρο ε, πληροφορίες, μάκρο στοιχεία για να συμπληρωθεί η εικόνα των στοιχείων της ΕΜΠΑ. Έτσι με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε να μην συμπεριλαμβάνουμε συστημική κίνδυνη στον υπολογισμό του προτύπου κινδύνου ώστε να συμπληρωθεί αυτό. Ευχαριστώ. Αν με επιτρέπετε να συμπληρώσω το ερώτημα του κ. Καμφά για το value at risk. σε όλα τα χρηματιστήρια, σε όλες τις αίθουσες συναλλαγών ε, και σε σχέση με τη χρήση του value at risk και την αξία που έχει σε περίπτωση κρίσης. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο. Ε, το είπε και η Κλάουτια Μπούχο ότι τα μοντέλα αυτά έχουν την αξία τους, είναι ευφύ, αλλά το θέμα είναι το εξή. Πρόκειται για μοντέλα τα οποία είναι χρήσιμα σε καιρό κρίσης. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το αστείο λοιπόν, που δεν είναι βέβαια και τόσο αστείο, τέλο πάντων παντού ακούγεται και θα το πω στα αγγλικά γιατί είναι η γλώσσα των χρηματοστριακών αγορών, Είπε ο κύριος Καμφέ ότι βασίζεται σε υποθέσεις, στατιστικών στοιχείων, ε, οι αποστάσεις και η κατανόμη λοιπά. Λοιπόν, ποιο είναι το αστείο τώρα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διέπονται από δύο πράγματα, το φόβο και την απληστία. Και αυτά ναι. δεν ακολουθούν τους νόμους ε, των, ε, της κατανομής. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί αυτό σε περίοδο κρίσης. Το ξέρουν όλοι οι ε, χρηματιστές αυτό δεν θέλουν εκείνη τη στιγμή έναν ε, ε, υπολογιστή που θα τους πει ποιος είναι, ποιος είναι ο κίνδυνος. Και τώρα περνάω σε πιο σοβαρά θέματα ή πιο τεχνικού χαρακτήρα. Αυτή μέθοδος, η κυρία Μπουχ ε, το ανέφερε, με τη διάσταση της συσχέτισης, το correlation, είναι ακριβώ η μέθοδος η οποία οδήγησε σε αυτό το, τριπλό α, αυτή την ε, ταξινόμηση, είδαμε τι έγινε το 2007-2008. Είπαν όλοι οι διαξιολόγοι, έχετε τριπλό α, μπορείτε να προχωρήσετε και τα λοιπά. Την ίδια μέθοδο αυτή την παίρνουμε και στο ΟΚΑ 4 Βασιλεία 3 ίδια αίτια παράγουν ε, ίδια συνέπειε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Ένα άλλο θέμα ε, προ τον κύριο Καφρά πάλι. Το ποιο είναι το πρώτο λιθαράκι αυτό. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, να μου επιτρέπετε. Δηλαδή, κάτι πολύ απλό είναι το πρώτο αυτό λιθαράκι που επιτρέπει να ελέγξουμε τι συμβαίνει και μετά φτάνουμε και στο δεύτερο λιθαράκι. Αλλά το πρώτο είναι ένα πολύ απλό μοχλό που μα επιτρέπει να δούμε πού πατάμε, πού πηγαίνουμε και τουλάχιστον κατά πόσον θα ξεφύγουν τα πράγματα ή όχι και να έχουμε μια σχέση μεταξύ ιδίων πόρων του κεφαλαίου που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι. Το προφανές, αλλά το θέλω να το επενδύσω σε σχέση με τον κίνδυνο. Και έπειτα δεν αρκεί ο μοχλός, γιατί όπως υπόθηκε και από τον κύριο Ενρία και από άλλους, είναι σημαντικό ο υπόπτης να είναι σε θέση να συζητήσει με μια τράπεζα, το είπε και η κυρία Γκραμπέρ, να μπορεί να πάει να συζητήσει με την τράπεζα, να αναλύσει τους κινδύνους, να συζητήσει, να πει ορίστε αυτός ο κίνδυνος είναι σημαντικός και η λογική ε, μιας ε, τέτοιας μοντελοποίησης θα μπορούσε να έχει νόημα. Βάζουμε πρώτα το μοχλό που είναι η μια ασφαλιστική δικλίδα και έπειτα χρησιμοποιούμε τα risk weights, δηλαδή τις σταθμίσεις κινδύνου για αυτό που είναι παρακολούθηση μέσω ελέγχου Παρακολούθηση. Αν βάλουμε τα risk weights στην αρχή, ουσιαστικά ε, δημιουργούμε μια μεθοδολογία που δεν λειτουργεί. Ε, δεν ξέρω να κατάλαβα πολύ καλά, αλλά το σύστημα το οποίο περιγράφεται, που ήταν και στις ΕΠΑ, leverage ratio, ένας ε, λόγος μόκλευσης που πραγματικά δεν απέτρεψε το αντίστοιχο μάλιστα την κρίση. Συμφωνώ μαζί σας ε, ότι σε περίπτωση κρίσης ε, οι σταθμίσεις κινδύνου πράγματι δεν μπορούν να προβλέψουν ή να, αναγγείλουν μια κρίση, αλλά στο 99,99% σε κανονικές συνθήκες οι τράπεζες και οι υπόπτε βοηθούνται από αυτό, από αυτές τις σταθμίσεις να υπολογίσουν το επίπεδο των κινδύνων. Με Briefly. Να απαντήσω, ναι. Να απαντήσω σύντομα, συμφωνώ απόλυτα ότι τα risk weights, οι σταθμίσει κινδύνου, είναι έτσι. Γι' αυτό και συνόψισα από την πρότασή μου στα εξή ότι αρχικά κάνουμε το leverage, που πρέπει να είναι απλό και αποτελεσματικό, όπω είπα, και επιπλέον να έχουμε αυτό το σύστημα risk weights, ώστε οι υπόλοιπε να μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των κινδύνων των τραπεζών για να αποφύγουν καταστάσεις τύπου Βασιλεία 1. Άρα όχι η Βασιλεία 1, είπαμε. Έχει κάποια λατώματα η Βασιλιά. 1. Είχαμε μείωση του, της μόχλευσης, αλλά μετά έχουμε τις, τον πειρασμό, αν θέλετε, τη τάση των τραπεζών ε, να ε, ξεφεύγουν λίγο σε διαφορά τη μόχλευση και τους ίδιους πόρους. Στη Βασιλεία 2 είπαμε κάνουμε το αντίθετο. Είχαμε ευρωπαϊκές τράπεζες με 30, 40, 50, 60. Τη μόχλευση ξέρουμε τι έγινε. Βασιλεία 3 γιατί όχι, ίσως θα μπορούσε να είναι η χρυσή τομή. Δηλαδή, ξεκινάμε με περιορισμό των σημαντικών κινδύνων που αναλαμβάνουν τράπεζες με την υπερβολική μόχλευση και έπειτα αφήνουμε στους επόπτες τη δυνατότητα να κάνουν το εποπτικό τους έργο, εποπτικό έργο που είναι σημαντική λέξη, και με τη μέθοδο risk weight των σταθμίσεων κινδύνου να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες για να ελέγχουν τον κίνδυνο, να είναι λογικός, στα όρια του λογικού. Αυτή λοιπόν η λογική της ΟΚΑ 4 και Βασιλεία 3 αντιστροφή για να μην φτάσουμε στη Βασιλεία 1 ξανά. το καταλάβαμε νομίζω αυτό. Ο Ανδρέα θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Ναι, καταλαβαίνω πως ε, βεβαίως ε, πάρα πολύ είναι υπέρ του λόγου μόχλευσης και δεν θέλω να τοποθετηθώ κατά. Είναι σημαντικό εργαλείο. Αλλά ε, θέλω να πω και ορισμένα άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο λόγος μου έχει μια σημαντική έλλειψη. Όταν πάμε σε μια κατάσταση όπου αυξάνονται οι κίνδυνοι και οι τράπεζες πλησιάζουν ε, η κατάστασή τους εν πάση περιπτώσει επιδεινώνεται, το κίνητρο για τους ε, διοικούντες είναι να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο, γιατί αυτό δεν φαίνεται. Οπότε το να περάσουν από στοιχεία χαμηλού κινδύνου σε στοιχεία υψηλού κινδύνου ε, δίνει τον ίδιο λόγο μόχλευσης, δίνει περισσότερο εισόδημα στην τράπεζα για να παίξουν αν θέλετε και έτσι υπάρχει και περισσότερο εισόδημα όπως είπαμε. Οπότε η ιδέα ότι υπάρχουν κάποια απλά μέτρα με τα οποία φεύγουμε τις κρίσεις είναι πάρα πολύ απλουστευτική. Τα απλά μέτρα δυστυχώς ε, αποτελούν ε, κάτι το οποίο εύκολα παρακάμπτεται όταν μιλάμε για την ε, καινοτομία στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε απλές απαιτήσει και μετά σε λίγες μήνες θα έχουν βρεθεί τρόποι να παρακαμφθούν αυτά. Οπότε αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι υποπτικές αρχές να μπορούν να μπουν στο πώς ε, διαχειρίζονται και μετράνε τον κίνδυνο τράψης και να είναι αρκετά σκληροί. Οπότε ο λόγος βεβαίως μόχλευσης ως γενικό μέτρο, αλλά πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να αντιληφθεί το πώς μετράνε τον κίνδυνο η εποπτική αρχή και να αυξήσουν τις απαιτήσει τους εάν δουν πως αναλαμβάνεται πάρα πολύ μεγάλο Ε, συμφωνώ πλήρως με τα επιχειρήματα που ακούστηκαν και από τον κυρία Καθηγήτρια και τον κύριο Φίλιππονα όσον αφορά τα μοντέλα. Έχω δει παραδείγματο χάρη στα stress test. Είδαμε πάρα πολύ περίπλοκες καταστάσεις. Ε, μιλάμε για εξισώσει στα μοντέλα που λειτουργούν κανονικά υπό ΚΣ, αλλά όταν μπούμε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι ακραίες οι αντιδράσεις και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ μοντέλων. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία να αντιδρούν πολύ γρήγορα και ακραία και άλλα μοντέλα τα οποία δεν μετακινούνται που είναι κάτι το άλλο για μας. Οπότε ο πλούτος των πληροφοριών που λαμβάνει η υποπτική αρχή δεν πρέπει να χάνεται. Πρέπει να έχουμε όλους τους μοχλούς αν θέλετε στη διάθεσή μας. Τέλος για τη διαφορετική ερμηνεία της ε, Οδηγίας Κεφαλαϊκών Απαιτήσεων 4. Είναι σημαντικό αυτό. Ήδη υπάρχουν κάποιοι τομείς ο οποίους μας ζητήθηκε να συνεργαστούμε με την Κοινή Επιτροπή. Π.χ. στα μέτρα τα κεφαλαιακά και βεβαίως τον ορισμό του κεφαλαίου στους δύο τομείς που πρέπει να είναι σωστός για να αποφύγουμε προβλήματα και στις δύο περιπτώσεις για να μην παρακαμφθούν τα κριτήρια σε έναν τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκη, έτσι. Ναι, έχω διάφορες ερωτήσεις για διάφορους. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Ενρία. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία είπατε, αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο και δεν θα ήθελα να λέτε διαφορετικά πράγματα εσείς από το Συμβούλιο Συστημική σταθερότητα. Ήρθε εδώ πέρα το πρωί ο κύριος Τρισέ και είπε ειδικά πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν ε, μακροπροληπτικά μέσα παραπάνω από αυτά τα οποία από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εγκαίρως. Και το ίδιο είπε και ο Ζακ Τελαροζιέρ, ότι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να πάνε παραπάνω. Εσείς είπατε πως η αύξηση βεβαίως ε, του κεφαλαίου είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε πάρα πολύ δύσκολα να γίνει. Θα ήθελα όμως ε, να συμφωνήστε εσείς με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτική Αρχή για το ποια μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πέρα από το υψηλότερο κεφάλαιο. Π.χ. στην Ιρλανδία θα έπρεπε να έχουμε υψηλότερη αξιολόγηση κινδύνου για τα δάνεια, για τα ακίνητα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή για να έχουν αυτή τη διακριτική ευκαιρία οι χώρες, αλλά έχουμε αυτή τη μέγιστη εναρμόνιση γιατί είναι ανησυχή ειδικά για χώρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους επιτόκια για να διαχειριστούν τον κίνδυνο δεύτερον. Η Erste Bank είναι πάρα πολύ σημαντική. Είστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειοδότης στην Ανατολική Ευρώπη και σε ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα όταν είχατε αυτές τις δύσκολες ανακοινώσεις χτες. Και συμφωνώ βεβαίω πράγματι για το ότι πρέπει να υπάρχει δανεισμό σε μικρές επιχειρήσεις και το πάθος που έχετε για το ότι ε, δεν, δεν βασίζεται συνεχώς στην ανασυσκευασία δανείων. Μιλήσατε βεβαίω για διαφάνεια ειδικά στον αφορά τα ομόλογα, αλλά απευθύνεται και μια έκκληση για την εφαρμογή της Βασιλείας 3 και να μην ζητάμε εξαιρέσεις και παρόλα αυτά η ομάδα σας ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα και ζήτησε εξαίρεση από το άρθρο 79. Ναι, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, όπως το ερμηνεύω εγώ, όπως ερμηνεύω εγώ αυτές τις εγγυήσεις που έχετε μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών σας, είναι πως μπορείτε να αντλήσετε αυτές τις εγγυήσεις από τις περιφερειακές τράπεζες για να καλύψετε απώλειες στην Αυστρία. Θα μπορούσατε να έχετε αντλήσει αυτά τα λεφτά για να καλύψετε τη χασούρα σας στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία αυτά που ανακοινώσατε χτες και θα μπορούσατε να έχετε κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να περάσετε στη διαδικασία της χρεοκοπία, αν είχατε αρκετό κεφάλαιο. Δεν θέλω να περάσω τώρα στο επιχείρημα του λόγου μόχλευσης. Χρειάζονται νομίζω και τα δύο εργαλεία. Αφήστε που εγώ θεωρώ πως επιστρέφουμε πίσω στην Βασιλεία, αλλά ε, εσείς που ασχολείστε με την πραγματική οικονομία, γιατί μιλάμε για δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Λίγες ερωτήσεις λοιπόν. Μπορείτε να μας προτείνετε έναν εύκολο τρόπο να ασχοληθούμε με τον ΕΜΗΡ και την οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων. Δεν είδατε, κάναμε πολύ αυστηρά τα πράγματα όσον αφορά τις υπόλοιπες εταιρείε. Οπότε υπάρχει ένας άλλος τρόπος μέτρησης. Ε, επίσης συμφωνούν όλοι πως ήταν πολύ φθηνό το κόστος ε, δανεισμού και κάποια από αυτά τα οποία είπατε μου λένε πως ε, όταν μιλάμε για πάνω από 100 μονάδες βάσης όταν είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια είναι πολλά λεφτά. Τι άλλο ζήτημα έπρεπε να εξετάζουμε πέρα από το κόστος της χρηματοδότησης, πώς θα κάνουμε καλύτερα αυτή την ανάλυση. Κάποιος συνάδελφος γελούσε όταν ε, ε, είπατε πως εξαρτάται από την απόδοση του κεφαλαίου όταν μιλάμε για χαμηλόδρυμόχληση. Είναι δύσκολο πράγματι, ένα περίπλοκο μοντέλο και πρέπει να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία. Και θα ήθελα να επίσης να καταλάβω εσείς και οι τελικοί χρήστε, ε, οι δανειστές, οι δανειοδοτούμενοι με συγχωρείτε, ήσασταν ενεργημένοι στην ε, διαβούλευση της Κομισιόν πριν μας δώσει αυτές τις προτάσεις. Νομίζω πως καλό είναι να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις αμέσως. Νομίζω κάποιες, ε, Αντρέα, απευθύνθηκαν σε εσάς και οι υπόλοιπες στην Έρστε Σας ευχαριστώ πολύ πολύ σύνθετο και περίπλοκο το θέμα. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν συντομότερο, παρότι είναι εκτενέ το θέμα. Πρώτον, δεν ήμουν παρόν να ακούσω τι την παρουσίαση του Jean-Claude Trichet σήμερα το πρωί, αλλά γενικά συμφωνώ με όλα όσα λέει. Και δεν θέλω να στείλω κάποιο μήνυμα να σηματοδοτήσω τίποτα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Θέλω να είναι σαφές, ως επόπτες πρέπει να έχουμε την ελαστικότητα για την αύξηση των buffers, των ε, ε μαξιλαριών, αλλά και θα πρέπει να δούμε και τους κινδύνους ε, συγκεκριμένα. Εκείνο το οποίο δεν βλέπω είναι αντίφαση ή αντίθεση σε σχέση με αυτή την προσέγγιση, με την ιδέα της ε, μέγιστης ε, εναρμόνισης. Ε, ήδη σήμερα για μια ενοποιημένη τέτοια κατάσταση για μια χώρα, για την Ιταλία για παράδειγμα, έχουμε κανόνες για την κεφαλαιακή απέτηση επάρκειας για μια τρέπεζα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα αύξησης αυτής, αυτών των προϋποθέσεων αν υπάρχει ειδικό κίνδυνος. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέπεια παντραπεζικά και σε, από χώρα σε χώρα πρέπει να έχουμε ελαστικότητα. Για παράδειγμα για μια χώρα που έχει μια φούσκα ακινήτων πρέπει να μπορεί να αυξάνεται ο κίνδυνος για την έκθεση σε τέτοιου είδους κινδύνους, κινδύνους, ενώ αυτό μπορεί να μην ισχύει για μια άλλη χώρα. Και αν έχουμε την ίδια φούσκα σε δύο χώρε, αυτό πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Διότι, όπω είδαμε υπερβολικά καλά, τα εξωτερικά στοιχεία διαφορετικών κρατών είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Χρειάζεται ελαστικότητα, αλλά χρειάζεται και κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνουν όλα αυτά και να λειτουργήσουν όλα αυτά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα όμω εκεί, πιστεύω, όσον αφορά τι μακροοικονομικέ απαιτήσει, ώστε να έχουμε το πλήρε φάσμα εύρο των μέσων και εργαλείων όπω απαιτείται για τα μακροοικονομικά ας το πούμε έτσι, ε, στο νέο αυτό τομέα και για την δημιουργία των μπάφες των ζωνών ασφάλειας και με την Συμφωνία Βασιλείας και μετά όσα έχετε εξετάσει εσείς και το Συμβούλιο για ε, την Οδηγία περί κεφαλαιακής επάρκειας, κεφαλαιακών απαιτήσεων, μέσω όλων αυτών έχουμε συγκεκριμένους τομείς. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς που πρέπει να, να επεκτείνουμε το εύρος των ε, δράσεών μας σε αυτούς. Και έτσι νομοθετικά θα πρέπει να δούμε αυτή την ανάγκη όπου ανακύπτει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας, παρακαλώ. Ανδρέα. Πολύ σωστό και απόλυτα σωστά αυτό αν αυτά τα οποία αναφέραμε δεν κόστιζαν επιπρόσθετο κεφάλαιο όσον αφορά την αναλογία ή το ποσοστό μόχλευσης. Αν, έχουμε, αν είχαμε πέσει κάτω από την αναγκαία αυτή αναλογία θα έπρεπε να αναπληρώσουμε, να ξαναγεμίσουμε τα κεφάλαιά μας από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας. Αυτό είναι στη συμφωνία μας και είναι ισχυρότερο στις συμβατικές αυτές υποχρεώσεις ε, όσον αφορά για παράδειγμα ε, τις ε, συμβατικές σχέσεις με κανονικούς μεριδιούχους ή κατόχους μετοχών. Και έχουμε λοιπόν και εξαιρέσεις σε περίπτωση που χρειαστεί. Αν αλλάξουμε για παράδειγμα το, την αναλογία για, καταθέσεων από 75% σε 25% ή ακόμα χαμηλότερα. Είναι μεγάλη βοήθεια για την, τον δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτό. Και αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για την μοχλική επίπτωση, την μόχλευση. Σκέφτηκε κανείς ποτέ την ανατροπή των πραγμάτων, την αντίστροφη κατάσταση. Δηλαδή στις τράπεζες να τους πει κανείς ότι πρέπει να κερδίσετε αυτή την μόχλευση και όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση αυτή, τόσο χαμηλότερη πρέπει να είναι η αναλογία κεφαλαϊκής επάρκειας. Δηλαδή, όσο λιγότερο φορτώνεται το φύλλο ισολογισμού σας και δεν υπάρχουν ε, επιπρόσθετοι κίνδυνοι, τότε θα είναι χαμηλότερη η κεφαλαιακή σας επάρκεια που θα απαιτείτε. Δηλαδή αυτό θα σημαίνει ότι οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν όσον αφορά το εμπόριο και άλλες τέτοιες συναλλαγές από πλευρά τους. Εκεί θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να κερδίσουν χρήματα. Θα ήταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε πολύ αν μπορούσε να γίνει. Δεν θέλω να επιβάλλω αυτή την άποψη σε εσά, αλλά νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε το ίδιο και στην επίλυση κρίσεων. Δεν ξέρω αν ο Ρίτσαρντ έχει να προσθέσει κάτι. Η Βίκη νομίζω ότι έκανε τρία ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Πρώτο, κατά πόσο υπάρχει εύκολη λύση στη διασύνδεση του ΕΜΗΡ και τη ΟΚΑ 4. Η απλή απάντηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απλή σχέση. Δηλαδή, οποιαδήποτε συναλλαγή ωφελείται από την ε, εξαίρεση μη χρηματοοικονομικό τελικό χρήστη, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με διακριτικό τρόπο υπό το πλαίσιο της ΟΚΑ4. Η ισοδύναμη δανειακή αξία του κεφαλαίου, δηλαδή το κεφάλαιο θα πρέπει να βασίζεται στην ισοδύναμη δανειακή αξία της έκθεσης στην συναλλαγή παραγόγων, ενώ αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερο αυτό, δεν ισχύει η ισοδυναμία και από ό,τι μου λένε για τεχνικούς λόγους είναι δύσκολο να δεχθεί το σύστημα κάτι τέτοιο. Τώρα, η λήψη αυτού Υπάρχουν και άλλοι τομεί. Είναι διπλή καταγραφή, το double counting, ε, δηλαδή ε, απατηλό και ε, λανθασμένο και στην ενοιολογική του σύλληψη και στο σχεδιασμό του. Διμερής έκθεση που αναγνωρίζεται στους υπολογισμούς του CVA. Δεν εκτίθεται η τράπεζα σε ένα παράγωγο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Και σε ό,τι Φορά την ΟΚΑ 4, αν κατάλαβα καλά κάθε παράγωγο δεν ε, έχει καθεστώς επισφαλούς ε, ε, συναλλαγής. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος ε, για την τράπεζα, αν είναι πολύ μικρότερος ή μεγαλύτερος. Ό,τι αφορά τα spreads, τα CD νομίζω ότι θα έχουμε ανεδική πίεση στα spreads ε, των ασφαλιστικών κινδύνου. Το βλέπουμε και στους υπολογισμού του ΣΥΒΙΑ. Ούτε βοηθάει, ούτε λογικό είναι. Δεν βοηθά τον τελικό χρήστη. Δεύτερο ερώτημα. Κόστος δανεισμού. Και αν υπάρχουν άλλες πτυχές που μας δημιουργούν ανησυχία. Σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού, είναι συντομία να πω ότι το αν είναι 20 ή 160 μονάδες βάσης, αυτό εμένα δεν με δημιουργεί πρόβλημα. Το θέμα είναι όσο μεγαλύτερο ο δανεισμό, τόσο λιγότερη δυνατότητα επενδύσεων. Και σίγουρα το κόστο κεφαλαίου επηρεάζει και διέπει τι επενδυτικέ αποφάσει. Άρα δεν πρέπει να καταστούμε όλο και πιο δύσκολε να τι επενδύσει, να το χρήμα κοστίζει όλο και περισσότερο. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έκανε μια ιστορική δημοσίευση τον Αύγουστο φέτο σε ένα έγγραφο που λέει ότι η συνολική παραγωγική παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, είδαν Καναδά και ΙΠΑ συγκεκριμένα, επηρεάζεται σημαντικά από αυξήσει του κόστου ε, χρηματοδότηση. Και το επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι υψηλό κόστο ε, δανεισμού κάνει λιγότερο βελτιστοποιημένε τι επενδυτικέ αποφάσει. Και το βλέπουμε ε, στα συμπεράσματα του Διεθνού Ταμείου. Άρα, όλο και λιγότερο καλέ θα είναι οι επενδυτικέ αποφάσει που λαμβάνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη αύξηση τη αναπόφευκτη στο κόστο δανεισμού. Βέβαια, μπορούμε να δεχθούμε ότι θα χρειάζεται να αυξηθεί το κόστο. Ελπίζουμε όμω να έχουν καταλάβει. Ε, να έχει καταλάβει ο κόσμο ότι αυτό που λέμε είναι ότι ο συστημικό κίνδυνο δεν προκαλείται από το μη χρηματοοικονομικό τελικό χρήστη. Άρα δεν πρέπει να τον τιμωρήσουμε ε, υπερβολικά τον μη χρηματοοικονομικό τελικό χρήστη, γιατί αυτό θα είναι κοντόφορο. Τρίτο ερώτημα, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε στις διαβουλεύσεις. Θα πρέπει να πω ότι και εγώ ε, ίσως έχω μία ε, σύγκρουση συμφερόντων. Θα είμαι σε μια πλατφόρμα στις Βρυξέλλες με ε, μια συνάδελφό σας εδώ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ τέλος πάντων. Ε, πάντως είδαμε ότι δεν ήθελε πάρα πολύ η Κομισιόν να ε, συζητήσει μαζί μας. Ε, στους μη ε, χρηματοοικονομικού τελικού χρήστες σε ό,τι αφορά ε, την ΟΚΑ 4 και λυπούμε γι' αυτό. Και είναι ένα δείγμα νομίζω τη μεγάλη επιρροή που ασκούν οι τράπεζες ως ε, μοχλιά σχέση πίεση. Και είναι προφανή η λόγη. Άρα μας έκλεισαν την πόρτα, πόρτα κατάμουτρα αλλά φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι ακριβώ εμεί και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να εισακουστούμε, έτσι να ακουστούμε σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευση. Σα ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα τρει-τέσσερι γύρου ερωτήσεων. Αλλά το είπα και πριν, αν απαντάτε όλοι σε όλε τι ερωτήσει, δεν φτάνει, δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. εσύ ο επόμενο. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου θερμά να ευχαριστήσω για το ότι βρήκατε το χρόνο και πάλι να έρθετε και να συζητήσετε μαζί μας και σας το λέω ειλικρινά. Μετά από τον πρώτο γύρο είχα ησυχάσει περισσότερο από τότε που είχε αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και μετά από τον πρώτο γύρο είχα την εντύπωση, είχα αποκομίσει την εντύπωση ότι από τον δόκτωρο οι εξελίξεις που σκιαγραφήθηκαν τον τελευταίο δύο ετών είναι αντικείμενο κοινή συνένεσης ως προς τότε, δηλαδή το αμφίσιμο εγχείρημα Βασιλείας 2 όπως το είδαμε πριν από δύο χρόνια όπως στην Ακρόαση είπαν πολλοί καθόλου δεν θέλουμε κάτι τέτοιο τώρα βρέθηκαν σε ένα επίπεδο μετά από τις πρώτες συζητήσεις του πρώτου γύρου που ουσιαστικά έλεγαν εντάξει θα το κάνουμε αυτό είναι και σωστό και σημαντικό και θα προχωρήσουμε. Και πρέπει κάποια πράγματα να ρυθμίσουμε και να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε. Τώρα ακούω ότι βρισκόμαστε στη μέση της νομοθετικής διαδικασίας και μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Την 1η Πρώτου 2013 θα πρέπει το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο, ο μηχανισμός αυτός να αρχίσει να μπορεί να λειτουργεί αν εγκρίνουμε εμείς και το δεχθούμε. Όμως στην Επιτροπή Βασιλείας και στη Λέσχη των 20 έχουν αποφασιστεί αυτά, έχουν εγκριθεί. Και ακούω παρεμβάσεις ότι αν δεν αλλάξουμε ε, κάτι, σαν αυτό και δεν δίνονται απαντήσεις, ε, τότε τι, να κάνουμε κάποια πειράματα, να πειραματιστούμε και μετά βήμα προς βήμα να εντάξουμε όλα αυτά στο νομοθετικό πλαίσιο. Ε, αυτά μου είναι ανεπαρκή και γενικόλογα, υπερβολικά γενικόλογα και ανεπαρκή σε συνδυασμό με τις ε, διαδικασίες και διεργασίες στις οποίες βρισκόμαστε. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Και εδώ πάλι πρόσεξα και άκουσα από τους εισηγητές και μετά από τον πρώτο γύρο είχα την εντύπωση ότι είναι 4-1 το αποτέλεσμα, η αναλογία 4-1. Από εσά μάλλον θέματα και προβλήματα αρχής άκουσα μέχρι το ότι θα καταστούν όλα δαπανηρότερα κτλ. Και άκουσα συγκεκριμένες προτάσεις υπό επιφυλάξεις τι θα μπορούσε ακόμα να γίνει και τι θα μπορούσαμε να κάναμε. Γι' αυτό στη δική μου παρέμβαση θα ήθελα να πω το εξή. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς αν το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο σε περιόδους κρίσης θα είναι επωφελές και θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επωφελώς και γι' αυτό συντάσσουμε αυτή την οδηγία αλλά και δρούμε όχι μόνο για περιόδους κρίσης και δεν είναι μόνο απαντήσεις για περιόδους κρίσεων που θέλουμε να έχουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι επωφελή και σε περιόδους μη κρίσης ή ομαλές περιόδους που καλύπτουν την πλειοψηφία των χρονικών διαστημάτων στα οποία δρούμε. Πρώτη μου ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτησή μου. και εν συντομία αναφέρθηκε αυτό, σύντομα αναφέρθηκε, το ε, περιθώριο της εθνικής παρέμβασης όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και τα περιθώρια buffers. Λέγεται ότι σε σχέση με τις εθνικές ανάγκες που θα υπάρχουν θα μπορούν να διαμορφωθούν αυτά τα πλαίσια. Όμως εμείς δημιουργούμε ουσιαστικά την ενιαία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά Μέχρι ποιου βαθμού θα μπορεί να προχωρεί η εθνική ελαστικότητα για τη διαμόρφωση αυτών των περιθωρίων χωρίς ε, να υποστηριχθεί ο ανταγωνισμός ε, και χωρίς η δραστηριότητα επιχειρήσεων σε διασυνοριακές ε, δράσεις και συναλλαγές να δυσχεραίνεται η δραστηριότητα τραπεζών. Διότι διαφορετικά σε κάθε χώρα θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια και στην ίδια επιχείρηση. Και πέρα από την έγκριση εθνικών εποπτικών αρχών δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο ώστε τα κεφάλαια να βρίσκονται εκτός ας το πω έτσι ορίου ε, που θα απαιτεί το αλλού ή για άλλους. Αυτό είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Η τρίτη ερώτηση αφορά ε, εσάς κύριε και εδώ αναφέρθηκε σε σχέση με την επιθυμία που εκφράστηκε όταν το ΕΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί, τότε θα πρέπει να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί η Βασιλεία 3 ως συμφωνία. Θα τα καταφέρετε μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι το 2000, δηλαδή 12 Ιούλιο να τα έχετε ολοκληρώσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις και διατάξεις. Θα τα καταφέρετε, διότι τον Ιούλιο 2012 εκπνέει, είναι η τελευταία καταληκτική προθεσμία για να τα εγκρίνετε όλα αυτά, αν θέλουμε την 1η Πρώτου 2013 να αρχίσουν να ισχύουν. Και ρωτώ με, διερωτώ με λοιπόν, είσαστε με τις 153 αυτές προτάσεις ή απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνοι ή δεν τις θεωρείτε μήπως και εσείς υπερβολικές και πολλές από αυτές περιτές. Θα πρέπει τότε να δουλέψουμε και να υπάρξει διάλογος για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Διότι κατεπηγόντως θα χρειάζεται κάποια τα θέματα του κανονισμού να ρυθμιστούν και να μην περιμένουμε το ΑΕΠΑ. Γι' αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε, να μου αποσαφηνίσετε αυτό μου το ερώτημα και η τελευταία μου παρατήρηση. Όλα περιστρέφονται γύρω από τη στάθμιση και αξιολόγηση. Αφενός στάθμιση και αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων. Θα ήθελα να ακούσω μια άποψη από πλευρά σας, μια πρόταση. Τι θα γίνει με αυτά τα ομόλογα. Και από την άλλη πλευρά την σημερινή χρονική στιγμή η αρνητική αξιολόγηση όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Αντρέα πώς θα καταλήξουμε λοιπόν σε triple A rating στην αξιολόγηση φερεγγιότητας τριπλού α για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα υπάρξει ισοδίκαιο πεδίο δραστηριοποίησης μεταξύ των μεν και των δε διότι υπάρχει κίνδυνος κάποιοι να έχουν σταθμιστεί ε, με ε, διαφορετικό τρόπο και να δυσχεραίνεται η ε, εμπλοκή τους και πώς θα καταλήξουμε στην αξιολόγηση των κεφαλαίων που θα μπορούσαν να, είναι, να δημιουργούν το μεγαλύτερο κίνδυνο και πώς μπορούμε να γυρίσουμε, να αντιστρέψουμε τα πράγματα σε σχέση με τα συγκοινωνούντα δοχεία και την αναλογία, τον λόγο που θα ισχύει για τα κεφάλαια που θα απαιτούνται για την κεφαλαιακή επάρκεια στα συγκοινωνούντα αυτά δοχεία. Αν γίνεται την ανάλυση σας με μια συγκεκριμένη πρόταση να την συμπληρώσετε. Οπότε, ποιος θα απαντήσει πρώτος. Ντομινίκ. Σε ό,τι μας αφορά ως μια μεγάλη τράπεζα, εμείς ποτέ το σχέδιο της Επιτροπής δεν το εννοήσαμε ως ένα σενάριο κρίσης, ιδίως ό,τι αφορά το κεφάλαιο. Μπορούμε να πούμε ότι οι επόπτες ε, επεξεργάζονται το θέμα εδώ και 20 χρόνια, ξέρουν τη δουλειά τους, επομένως υπάρχουν πράγματα τα οποία ίσως θα πρέπει να τα ξαναδούμε στο περιθώριο, αλλά νομίζω ότι γενικά το έχουμε αντιληφθεί ως κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε και δεν έχουμε πρόβλημα αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά την ρευστότητα, νομίζω ότι έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις μας για το ίδιο και η Κομισιόν, γιατί προβλέπει να υπάρχει μία περίοδο παρατήρησης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αντικυκλικές, τα αντικυκλικά μαξιλάρια, την αντικυκλική προστασία, πρέπει να γίνουν παραλλήλως ο κύριο Κάρας. Ένα πράγμα. Ένα σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη δική μας επιθυμία σε διαφοροποίηση με τη συμφωνία για την Συμφωνία Βασιλείου για την υποχρεωτική αξιολόγηση έκανε λόγο. Τώρα, άμα ακούσουμε τα όσα λέγονται σε αυτή τη συζήτηση, όπου η αναλογία αυτή παίρνει μεγαλύτερη σημασία για κάποιους από τους παρεμβαίνοντες προλαλήσαντες, από ότι ο άλλος πυλώνας, ε, τότε διαρωτώ βρισκόμαστε καν στην αξιολόγηση και μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο ή θα καθοριστεί η αναλογία αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε de facto να μην είναι αναλογία, ε, να μην είναι αξιολόγηση ή στάθμιση αλλά εφαρμογή της συμφωνίας αυτής κατευθείαν. Ευχαριστώ. Εσείς μιλάτε για τον πυλώνα 1 δηλαδή να εφαρμοστεί. Ε, Είχα πει ότι δεν λειτουργήσε καλά στη ΣΥΠΑ το εργαλείο αυτό, ούτε και στον Καναδά, που ήταν ε, οι δύο χώρες που εφάρμοσαν αυτό το εργαλείο. Δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση κρίση. Άρα, νομίζω ότι καλό είναι, τα είπα και πριν, μεταξύ του Τιερή και μου ε, υπάρχει ίσως μια απόσταση, αλλά Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για τους επόπτες. Μπορεί να δώσει κάποιες τάσεις σε σχέση με άλλα εργαλεία, αλλά θα πρέπει, πιστεύουμε, να μείνουμε σε αυτή την ε, προσέγγιση με τα weighted assets, risk weighted assets. Και αυτό θα πρέπει τα υπόλοιπα να τα δοκιμάσουμε με κάποιο τρόπο. Claudia, you want to come in, yes. Θέλετε εσείς να με Θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω τις τρεις ερωτήσεις σας. Η πρώτη. Ε, μιλάμε απλά για μια κατάσταση κρίσης με τις προτάσεις αυτές. Κοιτάξτε, το σκεπτικό είναι πως ε, το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο μειώνει τις επιπτώσεις της ε, κρίσης. Ότι δηλαδή η κρίση δεν είναι μόνο εξωγενείς παράγοντες, αλλά και το πώς κατανέμονται τα στοιχεία του, του ενεργητικού. Δηλαδή μιλάμε για πρόληψη της κρίσης. Τώρα το πώς η ευελιξία είναι αναγκαία. Είναι αναγκαίο να έχουμε κοινούς κανόνες ε, για το τι είναι μετοχικό κεφάλαιο κτλ. Αλλά Ακούστηκε επίσης το ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία για να λάβουμε υπόψη τις φούσκες ε, που σχηματίζονται σε συγκεκριμένες τομείς αγοράς. Οπότε πρέπει να πάμε κάπου πέρα από τα ελάχιστα. Αντιλαμβάνομαι αυτή την ανάγκη τώρα. Το ποια στάθμιση κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα με ρωτήσατε απευθείας. εξέφραξα βεβαίως την αντίληψή μου για το λόγο μόχλευσης και μετά βεβαίως η απάντηση είναι σαφής γιατί και τα κρατικά ομόλογα θα πρέπει βεβαίως να έχουν αντίκρισμα σε μετοχικό κεφάλαιο όπως οποιαδήποτε άλλη επένδυση της τράπεζας. Δεν έχω να σας πω κάποιο νούμερο για την στάθμιση του κινδύνου, αν αυτό θέλετε. Ναι. Νομίζω πως είναι κάπως αργά να περάσουμε σε αλλαγές τώρα. Στον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα γίνονταν εύκολα με κάποιες τεχνικές αλλαγές, δηλαδή απλά να, βελτιωθούν, να βελτιωθεί ο λόγος συσχετισμού στο πλαίσιο της Βασιλείας 3 για επιχειρήσεις με τίσιο τζίρο μέχρι, δεν ξέρω, 100 εκατομμύρια και να εισαχθεί όπως έγινε ήδη στη Βασιλεία 2 ένας λόγος εξορρόπησης για την λιανικό δανεισμό και νομίζω πως υπάρχουν αρκετά στατιστικά δεδομένα που μας λένε πως αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο που θα αντανακλά τον κίνδυνο των δανείων λιανικής του χαρτοφυλακίου αυτού και Τελευταίο θα ήταν να βελτιωθεί κάπως ο λόγος ε, ρευστότητας. Οπότε, αυτή τη στιγμή ο λόγος ε, των καταθέσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα 75%. Δεν ε, εκτοπτρίζει αυτό την σταθερό, την κατάσταση. Είναι πολύ πιο σταθερό πιο σταθερές αυτέ οι καταθέσεις και το να το μειώσουμε νομίζω το βοηθούσε πάρα πολύ και Βεβαίω από εκεί πέρα δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση όταν μιλάμε για τον λόγο μόχλευση. Υπάρχουν λοιπόν σαφή στοιχεία πόσο λόγο μόχλευση έχει πάει στον πυλώνα 2 και εκεί πρέπει να μείνει και δημιουργεί ε, σοβαρά προβλήματα και είναι ε, ένας ε, επιφανειακός λόγος, δεν τίθεται ζήτημα ο λόγος αυτός σταθμισμένων ε, στοιχείων είναι πράγματι πιο ουσιαστικός και τεχνικά καλύτερος. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό. Εάν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη για να δανείσει την πραγματική οικονομία και αντιστρέφουμε τον λόγο της μόχλευσης και λέμε στις τράπεζες πως πρέπει να κερδίσετε trading το οποίο κάνετε και τα ομόλογα μέσω δανεισμού στην πραγματική οικονομία, δηλαδή όσο περισσότερο δανείζετε στην πραγματική οικονομία, τόσο περισσότερο σας επιτρέπουμε να προσθέσετε και κάτι άλλο, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε παραπάνω γιατί μετά θα έχετε κύρια βασικά ίδια κεφάλαια που δεν θα είναι 8-9% αλλά θα σας βάλουμε ένα 25% εάν είναι ένα 10% του, του συλλογισμού σας και το υπόλοιπο είναι με χρεόγραφα οποιοδήποτε είδους. Νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να, να το σκεφτούμε. Οπότε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον δανεισμό είναι απλό και τεχνικό. Το άλλο ζήτημα όμως είναι κάπως σοβαρό εγχείρημα και πολλοί θα έχουν διαφορετική άποψη από αυτού. Μάλιστα. Ο Ρίτσαρντ ήθελε επίσης να παρέμβει. Ναι, σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε με τι παρατηρήσει του υπολείπου πάνελ. Νομίζω πω ο κύριο Κάρα κατά κάποιον τρόπο με ρωτούσε το εάν θα έπρεπε να αλλάξει η... το έργο που έχει γίνει από την Κομισιόν. Η απάντηση είναι όχι, γιατί έχουν δείξει κάποιοι ειδικοί πως μπορούμε να επιτύχουμε το σωστό αποτέλεσμα με κάποια συζήτηση για τους υπολογισμούς. Εάν μετανιώνω για κάτι είναι πως δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση καθώς ε, οι απαιτήσει, ε, οι προτάσεις ΟΚΑ έχουν φτάσει τώρα στη φάση που έχουν φτάσει. Ναι, σας ευχαριστώ. Να εξηγήσω κι εγώ πρώτα απ' όλα για να μην παρεξηγηθώ ε, με αυτά τα οποία λέω για την εθνική ευελιξία. Ο στόχος δεν είναι η οδηγία στόχο πρέπει να έχει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ομοιομορφία. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, ας δούμε τις... Ε, τα δικυκλικά αυτά μέσα προστασίας που νομίζω με σωστό τρόπο εισάγονται στην οδηγία. Υπάρχει λοιπόν ένα ενιαίο μέσο που ορίζεται στην νομοθεσία και μετά ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιείται βασίζεται σε κάποιες παραμέτρους, π.χ. απόκληση της ε, αύξησης ε, της πίστης μακροπρόθεσμα και βεβαίως ε, υπάρχει μια καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνδικού Κινδύνου και μετά γίνεται ένας έλεγχος ex για το πώς κάθε χώρα ενεργοποιεί αυτά τα μέτρα προστασίας για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Οπότε υπάρχει ένα μέσο που εισάγεται στην ομοθεσία, είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποιο μέτρο ευελιξία στα κράτη-μέλη για την ενεργοποίηση, γιατί βέβαια ο πιστοτικό κύκλο διαφέρει, αλλά υπάρχει ένα μηχανισμό που διασφαλίζει πω δεν υπάρχουν ασυνέπειε μεταξύ των χωρών. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέσα και βεβαίω, όπω ερμηνεύω εγώ την πρόταση τη Κομισιόν, επιτρέπεται να εισαχθούν και άλλα μακροπροληπτικά μέτρα. Δηλαδή, όταν μια χώρα, μια εθνική εκτιμιστική αρχή θεωρεί πω πρέπει να αυξηθούν οι απαιτήσει σε μια χώρα, πρέπει να πάει μέσω τη Κομισιόν. Και να ζητήσει την άδεια. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Θα ήθελα όμως να πω ε, όταν γίνει αυτό για μια χώρα πρέπει να ελέγξουμε το εάν χρειάζεται το ίδιο μέσο να εφαρμοστεί γενικά. Και ο ρόλος βεβαίως του νομοθέτη είναι να δει αν χρειάζεται κάτι τέτοιο και αν χρειάζονται αλλαγές στην νομοθεσία. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια συνέπεια. Υπάρχει μια ομοιόμορφη εφαρμογή. Τώρα, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, πράγματι είναι πολύ επίκαιρη η ερώτησή σας και εγώ ανησυχώ γιατί βλέπουμε πως δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις ε, πριν ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό από νομική σκοπιά. Αυτή είναι η άποψη της νομικής υπηρεσίας κομισιών. Αυτό όμως σημαίνει πως όταν αρχίσουμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε αφού ολοκληρωθεί η νομοθεσία δεν υπάρχει χρόνος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το τι κάνετε με το νομοθετικό κείμενο, εσείς και το Συμβούλιο, για να προσαρμόσουμε τις ε, προδιαγραφές μας σύμφωνα με τη συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα γύρω και βεβαίως πολύ το εκτιμώ αυτό. Τώρα για το λόγο μόχλευσης γρήγορα να πω πως η περίοδος παρατήρησης έχει μεγάλο ρόλο γιατί ο λόγος μόχλευσης στο παρελθόν δεν είχε επιτύχει γιατί ήταν ένα πολύ άμβλη μέσο και βασίζονταν μόνο στον ίδιο ισολογισμό. Τώρα η πρόταση στην ΟΚΑ είναι να αυξηθεί και να περιλαμβάνει δραστηριότητα εκτός ισολογισμού, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα, αλλά πρέπει βεβαίως να δούμε τη σωστή ρύθμιση, χρειάζεται μια περίοδος παρατήρησης για αυτό. Όσον αφορά τώρα το δανεισμό σε μικρομεσαίες επιχειρήσει. να σα πω πως λάβαμε επιστολή από τους επιτρόπους Μπαρνιέ και Ταγιάννη που μας ζήτησαν πέρα από τα όσα ανέφερα στις αρχικές μου δηλώσεις για το λόγο μόχλευσης να ελέγξουμε τον αντίκτυπο του νέου πλαισίου δανεισμού στις ΜΜΕ και να δούμε αν υπάρχει μια δυνατότητα ελάφρυνσης μέσω της μείωσης ε, της στάθμισης του κινδύνου ή της διεύρυνσης του κατοφλίου ε, των ΜΜΕ που είναι επιλέξιμες για το χαρτοφυλάκι αυτό και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σβέν. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω και να δώσω μια πιο ζωντανή ε, εντύπωση στη συνεδρίαση. Ξεκινήσαμε με τις ε, παρεμβάσεις ε, για τις ε, τραπεζικές ρυθμίσεις. Δεν ξέραμε ακόμα ότι έχουμε και συμφωνία όσον αφορά τη διαφάνεια και τα λόμπις. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος ε, έχω δύο σημαντικά ερωτήματα, δύο σοβαρά ερωτήματα πέρα από τα ανέκδοτα. Ε, η συζήτηση επί της ουσίας διεξάγεται για το αν θα υπάρξει μείωση ή αύξηση. Η σημαντική αύξηση στο κόστος ε, για το δανεισμό για την πραγματική οικονομία ή όχι. Κάποιοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι, άλλοι ίσως. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εμπειρικά δεν είναι, πρέπει να, να το δείξει η ίδια η πείρα. Είναι μια σύγχυση που δημιουργείται. Κατανότα ως ανέφερε ο Όρμαρ Κάρας Έχουμε μια παρουσίαση, μια εκπομπή στην τηλεόραση όπου Πάντα διαφωνούν στις συζητήσεις οι ομιλούντες, ε, είναι πολιτικοί όχι επιστήμονες. Μετά υπάρχει μια δοκιμή, μια ε, άσκηση στο ε, διαδίκτυο για αυτές τις παρεμβάσεις. Σας ζητώ λοιπόν να μας στείλετε εσείς τις εντυπώσεις σας ή τις απαιτήσει σας και θα έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε στην συνέχεια. Γιατί αυτά θα είναι τα ερωτήματα τα οποία ερωτούν οι πολίτες. Να δούμε τι λέτε εσείς. Σας καλούμε λοιπόν να κάνετε αυτό το εγχείρημα ως άσκηση και προσκαλούμε τον καθηγητή να μας δώσει κάποια στοιχεία, περαιτέρω στοιχεία, υπό το εμπειρικό πρίσμα της ε, ίδιας της εμπειρικής προσέγγισης. Ένα επιχείρημα με το οποίο ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι η αναλογία μόχλευσης, ε, ratio. Και εδώ για κάποιες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που έχουν χαμηλό ποσοστό κερδοφορίας και που λειτουργούν με μικρά περιθώρια, στενά περιθώρια. Διαρωτώ με, όταν λέτε ότι είσαστε υπέρ ε, μια τέτοια αναλογία ε, ε, ενό τέτοιου λόγου μόχλευση ή υψηλότερη μόχλευση όπω είπατε, αυτό θα είναι επιζήμιο για αυτή την προσέγγιση την τραπεζική για αυτέ τι επιχειρήσει που σε, σε κάποιου τομεί θα είχαμε το θέμα για παράδειγμα του δανεισμού που είναι κρίσιμο. Και η τελευταία παρατήρηση προς εμάς, διότι αντιμετωπίζουμε στη Γερμανία συχνά επιχειρήματα από μικρότερες τράπεζες που λένε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως τις μικρότερες και θα πρέπει να υπάρχει μια γενική εξαίρεση. Πώς το προσεγγίζετε εσείς υπό το πρίσμα σας. Θα έχουμε την ίδια αυτή προσέγγιση για τις τράπεζες όπως ζητείτε. Δηλαδή υπό τον τίτλο της, ε, του, ταμιευτηρίου θα υπάρχει η ένταξη στην κατηγορία όπως των άλλων τραπεζών τι γίνεται σε σχέση με τα πρότυπα υπό αυτή την προσέγγιση. Πού θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση και πού όχι. Ώστε οι σκληροί κανόνες να μην χτυπούν, να μην πλήττουν τους μικρούς που δεν είναι ικανοί να συμμορφωθούν αλλά θα εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Μόνο εγώ έχω απομείνει για να κάνω ερωτήσεις. Ε, θα ε, το κάνω τώρα και μετά θα μπορέσετε όλοι οι ομιλητές ε, να εκφραστείτε. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπε ο Ανδρέας, για παράδειγμα, για τη ρευστότητα και την διαφοροποίηση. Είναι κάτι το οποίο με προβλημάτιζε εδώ και καιρό και ιδίως όταν είδαμε επαναλήψεις στα CCP, στη Solvency 2, τη Φαγκαιρότητα 2. Για το, ε, και για το δημόσιο χρέος. Επομένως, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και άλλοι φορείς να ξεκινήσουν ίσως την επέκταση του καταλόγου, τη διεύρυνση του καταλόγου των πραγμάτων που πιστεύουν ότι μπορούν να τυποποιηθούν. Παραδείγματο χάρη τα covered bonds, αυτά τα ομόλογα μπορούμε να τα τυποποιήσουμε και ίσως αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και στα άλλα αξιόγραφα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μη εισηγμένες μικρές ε, εταιρείε χρησιμοποίησαν τα CLOs ε, πολύ πρόλες από αυτές. Και αυτές οι, ε, αυτοί οι τίτλοι ε, λίγουν όπου να είναι και δεν ξέρουμε αν θα αντικατασταθούν. Δεν ξέρω αν κάποιο σκέφτηκε μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούσαμε να πετύχουμε να υπάρξει το rollover αυτών των τίτλων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάθμιση κινδύνου, μας απασχολεί και μας εδώ 19 μήνες, 18 μήνες πρωτοψηφίσαμε στην Επιτροπή μας ένα ψήφισμα που αναγνωρίζαμε την ανάγκη ενδεχομένως να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των ε, διαφόρων. Ε, και είπαμε, είπε η Κλόντια για αυτό το μόχλο, μάλλον αυτό τον ε, λόγο μόχλι, Σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικά ε, τα γερμανικά από τα ελληνικά ομόλογα. Τελικά, πώς προσαρμόζουμε τις σταθμίσεις κινδύνου. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ το θέμα των ασφαλιστρών κινδύνων. Θα μπορούσατε ίσως να προβλέψετε κάποια καθεστώτα ευρύτερης έκθεσης δηλαδή να μπορεί να σχετίζεται με, τις με το μέγεθος της χώρας και να δούμε εκεί ποια θα μπορούσαν τα επιτόκια και τα spreads. Ο Τιερή επίσης είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τα παράγωγα και τις σταθμίσεις κινδύνου. Διερωτώ με, μήπως έχει δοθεί πάρα πολύ προσοχή, υπερβολικά πολύ ε, προσοχή ε, στην νομοθεσία για το hedging Ενθαρρύνουμε δηλαδή το hedging με τεχνητά μέσα. Αντί να βλέπουμε την, την, την πιθανότητα διαφοροποίησης, να έχουμε δηλαδή ένα ισοδύναμο hedging με επένδυση στην πραγματική οικονομία. Επειδή φιλελεύθερη δεν είμαι πολύ υπέρ του αποκλεισμού, της απαγόρευσης κάποιων πραγμάτων, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια προνομιακή στάθμιση κινδύνου προς την άλλη πλευρά. Diversity μου για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να το θαρρύνουμε, έστω και σε μικρή κλίμακα, και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις. Και ούτω καθεξής. Τελικοί χρήστες. Ο Κα Εμίρ. Είμαι και στους δύο τριμερείς διαλόγους, παρακολουθώ λοιπόν τα θέματα αυτά. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα που να έχει μια λογική. Σε ό,τι αφορά το trade finance, ε, νομίζω το ανέφερε ο Ρίτσαρτ. Και εγώ διερωτώ με αν είναι στη σωστή κατηγορία. Που υπάρχουν κάποιοι ιστορικού χαρακτήρα κατηγοριοποιήσεις. Μήπως ε, για να μην μακρηγορήσω επειδή βήχω και πνίγομαι, Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε όλους τους ομιλητές για να απαντήσουν. Έχετε να απαντήσετε και στα δικά μου ερωτήματα και στα ερωτήματα του Σβέν. Okay, Jerry, Λοιπόν, Τιερή, θέλετε εσείς να απαντήσετε πρώτα. Ναι, αρκετά σημεία. Πρώτα απ' όλα. Νομίζω πως δύο από τις ερωτήσεις του Σβέν έφυγε. Θα απαντήσω ούτως ή άλλως. Ε, σχετίζονται. Μίλησε για το κόστος δανεισμού θα ήθελα να επισημάνω το ότι υπάρχουν μελέτες από ιδρύματα σοβαρά όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, Δουνοτού, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, το Ινστιτούτο Max Planck, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, που μιλάνε για μηδενικό έως πολύ μικρό κόστος τραπεζικού δανεισμού, αλλά θα θα συντάξουμε και ένα έγγραφο να το τεκμηριώσουμε. Αλλά το, κόστο, το ζήτημα του κόστου δανεισμού, που όπω καταλάβατε εγώ θεωρώ πω είναι μηδέν έω αμεληταίο, είναι το ίδιο ε, ερώτημα που έθεσε ο Σβέν για τον λόγο μόχλευση. Δηλαδή, αν ο λόγο μόχλευση εμποδίζει την δυνατότητα χρηματοδότηση τη πραγματικής οικονομίας. Είμαι απολύτω πεπισμένο πω αυτή τη στιγμή πούμε πω περισσότερο μετοχικό κεφάλαιο δεν αυξάνει τον σταθμισμένο κίνδυνο των τραπεζών και άρα δεν αυξάνει τον κίνδυνο δανεισμού, δεν, αυξα... δεν επηρεάζει και τον δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Αυτό στο οποίο επιδρά και το είπαν πολλοί είναι πως ο δανεισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει μεγαλύτερη στάθμιση κινδύνου από ότι ο δανεισμός σε ένα κράτος. Αυτό έχει αντίκτυπο. Είναι πράγματι πιο επικίνδυνο για μια τοπική τράπεζα που ξέρει τον πελάτη της πολύ καλά να δανείσει Εάν ο κανονισμό λέει «Α, είναι πολύ πιο επικίνδυνο», τότε αυτόν έχει αντίκτυπο. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπατε και εσείς, Σάρων, για την ποικιλία στο hedging. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά. Ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε είναι η ποικιλία. Ο βασικός κίνδυνος είναι να έχουν όλοι τα ίδια πράγματα στα χέρια τους, να έχουν επενδύσει και να αποεπενδύουν την ίδια στιγμή γιατί έτσι δημιουργείται ένας παύλος κύκλος. Η καλύτερη προστασία είναι η ποικιλομορφία. Γι' αυτό εάν βάλουμε τη στάθμιση κινδύνου στην πρώτη γραμμή θα αρνούμε τους πάντες να έχουν τα ίδια να κάνουν τις ίδιες τοποθετήσεις και άρα αυξάνεται ο συστημικός κίνδυνος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ σοβαρό. Η προστασία λοιπόν όπως σας είπα, είναι μια τοπική λύση, όχι παγκόσμια. Τοπική λύση για το χύψη ίδρυμα. Η γενική λύση είναι αν υπάρχει ένα σύστημα με αρκετή ποικιλομορφία. Ναι, ναι, βεβαίω. Μιλήστε εσείς. Ναι. Ως καλή πανεπιστημιακός έχω κάποιες παραπομπές στις σημειώσεις μου, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, Βεβαίως υπάρχουν εμπειρικέ μελέτες που έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά θα διαβάσω εγώ τα, στοιχεία όπως αναφέρθηκαν. Πως το κόστος ε, δανεισμού είναι σχετικά μικρό σε αυτές τις μελέτες και ε, βεβαίω ανεξαρτήτως του κόστους που υπολογίζουμε πρέπει να το συγκρίνουμε με το κόστος της κρίσης και τότε βεβαίω η ανάλυση είναι ξεκάθαρη. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ανέφερα. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε την ρύθμιση των τραπεζών με το να λύνει άλλα προβλήματα που έχουμε αλλού στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και αλλού έχουμε προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε αλλά δεν είναι εδώ πέρα ο τόπος ε, η ρύθμιση δηλαδή των τραπεζών να γίνει λιγότερο άκαμπτη για να λύσουμε προβλήματα αλλού. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε, προκύπτει συχνά είναι το τι συμβαίνει με τον κίνδυνο των τραπεζών εάν αυξηθεί ο λόγος ε, κεφαλαιοποίησης. Και εκεί πέρα η ερμηνεία που κάνω εγώ είναι πως η ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες θα μειώνονταν γιατί υπάρχει λιγότερο κίνητρο ή δυνατότητα να μετακυλιστεί ο κίνδυνος αυτό στην κοινωνία. Αν δείτε ιστορικά το τι γίνεται θα δείτε πως τα επίπεδα του μετοχικού κεφαλαίου ήταν πολύ υψηλότερα αλλά και ο κίνδυνος που είχαν οι ιδιοκτήτες αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερος γιατί υπήρχε και κάποιο είδου δίκτυο ασφαλείας για τις τράπεζες οπότε θα μπορούσε η ανάληψη αυτού του κινδύνου να μειωθεί με υψηλότερο λόγω κεφαλαιοποίησης, αλλά βεβαίω μιλήσετε και για τους κανόνες της μεγάλης έκθεσης, κάτι το οποίο έχουμε στους γερμανικούς ε, κανόνες ε, ρύθμισης των τραπεζών, δεν ξέρω τι γίνεται αρκετά σε άλλες χώρες, αλλά οι υψηλότερε κεφαλιακές απαιτήσει δεν είναι πανάκια που λύνουν όλα τα προβλήματα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Δεν μπορούσε να είναι αυτός ένας τρόπο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να στραφώ στο θέμα ως ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρότερες τράπεζες στην τράπεζα ώστε να μην χρειάζεται να εφαρμοστεί η Βασιλεία 3 ή το CDR 4. Θα το ήθελαν ιδιαίτερα να υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις στα ταμιευτήρια, για παράδειγμα. Η απάντηση είναι απόλυτα ένα κάθετο όχι. Αν έχουμε ένα κανόνα κανονισμό στην Ευρώπη πρέπει να ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεν μπορεί να υπεκφύγει κανείς ένα κανόνα κεφαλαιοποίησης επειδή είναι μικρός. Και όπως ε, επισημάθηκε, η συσσόρευση 500 μικρών τραπεζών μπορεί να είναι εξίσου συστημικός κίνδυνος όσο ο κίνδυνος που απορρέει από μια πολύ μεγάλη τράπεζα. Εξαιρέσεις θα ήταν κάτι παράλογο. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες ε, σε σχέση με ξεχωριστή αντιμετώπιση όσο αφορά τις μεγάλες τράπεζες επειδή ουσιαστικά χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία παίρνουν ε, καταθέσεις ε, από τις αποταμιεύσεις των πελατών τους και χρηματοδοτούν εταιρείες, μικρές εταιρείες. Αν έχουν τέτοιου είδους αποθέματα μπορούν να επενδύουν σε κρατικά ομόλογα διότι θεωρείται ότι είναι τα λιγότερο επικίνδυνα ως επένδυση σε σχέση με άλλες επενδύσεις όταν έχουμε ε, ε, την αναλογία σε σχέση με τα αποθέματα μιας τράπεζας ε, και όταν βλέπουμε τώρα ότι ε, σε σχέση με τις καταθέσεις όταν υπάρχει μια χαμηλή αναλογία, έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση όσον αφορά το κρατικό χρέος, που είναι ένα συστημικός κίνδυνος αφέ αυτού. Το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή αποταμιευτική τράπεζα στην Δημοκρατία της Τσεχίας, που έχει πολλές επενδύσεις όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα της Τσεχίας, θεωρείται χωρίς κίνδυνο μόνο στην Τσεχία, όχι εκτός Τσεχίας. Και αυτό μας θέτει ενώπιον του γεγονότος που μάθαμε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια πρόσφατα ότι αυτό είναι κίνδυνος. <clears throat> Το, ε, η ε, οδηγία περικεφαλαιακών απαιτήσεων ε, αυτό προβλέπει. Το CRD4 δεν επιλύει το πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι άσχετα ό,τι και να κάνει κανείς, <clears throat> η Ευρώπη ως Ήπειρος με ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ε, ε, ομολόγων έχει πλέον ε, πάψει να υπάρχει. Δεν μπορεί αυτό να γυρίσει πίσω με την Βασιλεία 4. Γι' αυτό πρέπει αυτό, αυτή την κατάσταση να συμπεριλάβουμε στις ρυθμίσεις και στους κανονισμούς. Κανείς δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει τον κίνδυνο κακής διακυβέρνησης ή των επιπτώσεων κακής διακυβέρνησης εκτός ε, μιας συγκεκριμένης χώρας. Και αυτό είναι κίνδυνος και για συγκεκριμένες τράπεζες. Πρέπει να το δούμε. Μια μικρή τράπεζα στην Πορτογαλία μπορεί να έχει εξαιρετικό ισολογισμό. Εξαιρετικό ισολογισμό. Όταν όμως ε, η ρευστότητα αυτή είναι σε κρατικά ομόλογα της Πορτογαλίας, κανένας δεν την πάρει στα σοβαρά. Δεν θα είναι φερέγγια. Ευχαριστώ. then I'll come back to Richard and then... και μετά αυτό το παρατηρούμε είναι ότι το κόστος κεφαλαίου για τις τράπεζες αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά. Το κόστος ε, του συν 1% κεφαλαίου αυξάνεται όσο μειώνεται η αξία των τραπεζών. Αυτό σας εξηγούσα και πριν. Η λύση θα ήταν να μειωθεί ο παρονομαστής. Το ενεργητικό δηλαδή. Εν γέννη, συνεχίζει το δανεισμό προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, θα ήθελα να πω κάτι ακόμη. Στο παλαιό περιβάλλον, το ασφάλιστρο, το premium που έδιναν οι τράπεζε, μάλλον που όριζαν οι ευρωπαϊκέ τράπεζε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ήταν πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των αμερικανικών τραπεζών. Ήταν ένα οικοσύστημα, αν θέλετε, το οποίο λειτουργούσε με πολύ ε, πιο μικρό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, πολύ ευνοϊκότερο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και μάλλον το νέο σύστημα θα τα αλλάξει όλα αυτά. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η λύση θα είναι σιγά σιγά να πάνε τα πράγματα όπως και στις ΗΠΑ, αλλά σιγά σιγά, γιατί προς το παρόν δεν έχουν πρόσβαση στις κεφαλαγορές ή πολύ λίγη ε, πρόσβαση γιατί αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις με πολύ, γρήγορα, ε, πολύ γρήγορο δυναμικό ανάπτυξης, δεν αφορά αυτό όλες τις επιχειρήσεις επομένω. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς το πλαίσιο της ε, περίοδου παρατήρησης ε, για τον δίκτυ ρευστότητας, για το λόγο ρευστότητας, όλα αυτά θα αναλυθούν, θα δοκιμαστούν με πάρα πολύ λεπτομεριακό και αναλυτικό τρόπο, γιατί η ΜΜΕ, η χρηματοδότησή τους θα παραμείνει στο επίκεντρο ε, των προβλημάτων για τα επόμενα χρόνια. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο, μάλλον αν θέλετε, μια εξέλιξη η οποία θα είναι μακροχρόνια. Ευχαριστώ πολύ, ο Ρίτσαρντ. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για το κόστος κεφαλαίου. Όλοι θα χαιρόντουσαν αν λέγαμε ότι δεν θα υπήρχαν επιπτώσεις. Όμως είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί όταν έχουμε τον πρώτο κανόνα χρηματοδότησης ότι ε, έχουμε τις μεγαλύτερες αμοιβέ ε, και α, τη μεγαλύτερη ανταπόδοση με το ε, higher equity capital και αυτό θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη το κόστος δανεισμού για την πραγματική οικονομία Εν πάση περιπτώσει όμως, ε, ίσως ε, εδώ σε αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση. Για το θέμα του hedging δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω απόλυτα αυτή τη σκέψη σας, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να περιορίσουν τους κινδύνους όσο γίνεται, ώστε να αναχαιτιστούν, να μειωθούν οι κίνδυνοι σε σχέση με τέτοιου είδους συναλλαγές. Παράδειγμα, όταν έχει κανείς ε, συναλλαγές σε σχέση με πρώτες ύλες, ε, ο στόχος είναι να μπορέσει κανείς να θέσει περιορισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι στην πραγματική οικονομία για τους δείκτες για αυτού του είδους ε, τα, τις συναλλαγές ε, που δεν είναι ιδιαίτερα ε, θελκτικοί λόγω της έκθεσης στον κίνδυνο που είναι υψηλός και για την χρηματοδότηση. Συμφωνώ εν τα προβλήματα με την χρηματοδότηση όσον αφορά το εμπόριο με τις προτάσεις CRD4 και Βασιλείας 3 βρίσκονται στην απουσία πιθανότητας ε, να μπορεί να υπάρχει κάποια έκθεση σε κίνδυνο όσον αφορά τους ισολογισμούς ε, που να μην έχει ληφθεί υπόψη. Αυτό δεν αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή από τις προτάσεις, δεν μπορεί να ποσοστοποιηθεί. Και δεύτερον, όσον αφορά την ροή οριμοποίησης, οριμότητας, είναι ενός έτους και όχι λιγότερο από ένα έτος. Και πολλές τέτοιες συναλλαγές ε, έχουν μια πολύ μικρότερη διάρκεια χρονική και θα πρέπει να δούμε την ε, συνιστόσα της μείωσης ε, κινδύνου όσον αφορά τη διαφορετική χρονική περίοδο σε έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους. Σας ευχαριστώ για το θέμα της επίπτωσης όσον αφορά τον δανεισμό και δανεισμό για την οικονομία γενικά. Δεν είμαι πανεπιστημιακός, όμως πιστεύω ότι τα θέματα αυτά είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, πανεπιστημιακούς είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί ή να αναγνωριστεί αυτό. Είδα εμπειρικές μελέτες και πολύ καλές τέτοιες μελέτες που στοχεύουν ή δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Για μένα το σημείο το οποίο είναι σαφές είναι ότι εμπειρικά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν βλέπει κανείς ή θεωρεί ότι οι απαιτήσει κεφαλαίου είναι υπερβολικά χαμηλές, επειδή τώρα για παράδειγμα οι αγορές έχουν έκθεση στο κρατικό χρέος και τους κινδύνους ε, του κρατικού χρέους, της κρατικής υπεχρέωσης. Απλά έχουμε τόσο μεγάλες δυσκολίες ε, όσον αφορά χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων και το κόστος του χρήματος για αυτή τη χρηματοδότηση είναι τόσο υψηλό που πρέπει κανείς υποχρεωτικά χρησιμοποιήσει μόχλευση. Το να έχει λοιπόν κανείς κεφαλαϊκές απαιτήσεις που θα είναι αξιόπιστες, που θα είναι καλά υπολογισμένες και σταθμισμένες και θα είναι ισχυρές και θα προστατεύουν, ας το πω έτσι, από πλευρά ασφάλεια ε, του ε, μετόχου μια τράπεζα είναι θεμελιώδου σημασία για τη σωστή χρηματοδότηση. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να επιτευχθεί ο δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη πραγματική οικονομία. Ο μείζον κίνδυνο είναι ότι συμπιέζεται τόσο πολύ όσον αφορά το δανεισμό η πραγματική οικονομία και ο δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επειδή υπάρχει εντύπωση ότι δεν έχουν καλώ υπολογιστεί όλα αυτά τα πράγματα και οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι αξιόπιστο και επαρκώς ισχυρό και έτσι να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να βοηθήσουμε να μην είναι υψηλό πλέον το κόστος ε, χρηματοδότησης. Αυτή πρέπει να είναι η σωστή, α το πω έτσι, πορεία όσον αφορά την αξιολόγηση των πραγμάτων. Για την ρευστότητα, φερεγγιότητα και διαφοροποίηση όσον αφορά τον διαφορετικό εστιασμό, κατανοώ απόλυτα την παρατήρηση. Η Επιτροπή της Βασιλείας ξεκίνησε από την ιδέα ότι θα έπρεπε να έχουμε υψηλής ποιότητας ρευστά περιθώρια, περιθώρια ρευστότητας ως buffers, ως ε, δηλαδή μαξιλάρια ή αποσβέστες ε, κραδασμών. Για να... Πρέπει όμως να δούμε και την ανάγκη ύπαρξης μιας ε, ελαστικότητας, μιας ευληγησίας στη διάθεση κεφαλαίων δανεισμού και θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ομόλογα, για παράδειγμα, ενός κράτους και μετοχές και από πλευράς των ε, ε, εποπτικών αρχών που έδωσαν όθηση προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε πιο πέρα από τις αρχικές προτάσεις. Τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε πάλι αυτό το πλαίσιο. Να αναθεωρήσουμε να δούμε η σύνθεση, ε, η σύσταση είναι σωστή, δεν χρειάζεται περισσότερη πολυμορφοποίηση μεγαλύτερη ποικιλότητα όσον αφορά για παράδειγμα και την, το μείγμα με τις με τα, κεφαλ, κεφάλαια ή τα ίδια κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει πάλι κάτι να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να ρυθμίσουμε αυτούς τους τομείς. Να τονίσω επίσης ότι υπό συγκεκριμένο πρίσμα ήδη έχουμε αλλαγές υπό την Βασιλεία 3 όσον αφορά τις ε, αλλαγές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο δεσμός που θα υπάρχει θα είναι σε σχέση με άτομο προς άτομο ή αγορά προς αγορά. Τώρα, όσον αφορά για, τις, ε, για τα ομόλογα, ως εποπτική αρχή διαρωτάται κανείς, είναι σωστό να ζητά κανείς από τις τράπεζες να έχουν ε, ένα περιθώριο ε, για την απόσβεση κραδασμών όσον αφορά τα προβλήματα στις αγορές και πώς θα μπορούσε να υπάρξει η αναγκαία οριμότητα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά χωρίς να υπάρχει ε, κάποια αντίφαση ή αντίθεση έκδηλη. Και πάλι εδώ πρέπει να δούμε το θέμα του κρατικού χρέους, για το hedging και τα hedge funds. Συμφωνώ υπό το πρίσμα του ότι εδώ υπάρχει ένας τομέας όπου μάλλον υπάρχει εδώ υπό την ε, μακροοικονομική ε, προοπτική ε, για το δανεισμό μια αντίφαση ή μια αντίθεση. Όμως ως επόπτης, εποπτική αρχή πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει μικρότερος κίνδυνος θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι θα πρέπει να δούμε το πώς μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ή όχι. Και η SRB θα έπρεπε να αναλάβει έργο σε αυτό το τομέα, να δραστηριοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύνοψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που ήρθατε. Έχουμε ακόμα άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη το στο οποίο είναι η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιριών. Θα φύγω εγώ και θα αναλάβουν μια αντιπρόεδροι για την ώρα που έχει μείνει. colleagues, can, can I ask you to... Uh, to... Λίγο ήρεμα παρακαλώ να εκενώσετε την αίθουσα γιατί ο χρόνος είναι λίγος για το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Τάισεν, η συγγητριά μας είναι εδώ. Sorry, you, you need to leave and have your conversations outside. Ε, Περάστε έξω για τις συζητήσεις, αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και να σεβαστούμε και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 Κύριε Κυρία Τάισεν, έχετε τον λόγο για να παρουσιάσετε την πρότασή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν αν δεν το διαβάσατε, να σας διαφωτίσω λίγο γρήγορα. Αυτό το οποίο λάβαμε είναι ένα κοινό σετ ευρωπαϊκών κανόνων για τον υπολογισμό φορολογικής βάσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Είναι μια πρόταση, ένα σύστημα ε, που μας οδηγεί σε ένα σύστημα εθελοντικό. Αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα ενιαίο κοινωνικό σύστημα. Δεν θα είναι υποχρεωτικό. Θα έχουμε δηλαδή ένα 28ο σύστημα φορολογίας εταιριών, αλλά όταν το επιλέγει μία εταιρεία, αυτομάτως θα μπορεί όλες τις συναλλαγές της να τις δηλώνει με βάση αυτό το ένα σύστημα και μπορεί άρα να περιοριστεί σε μία δήλωση και να έχει να κάνει με μία φορολογική διοίκηση. Την κύρια λεγόμενη φορολογική διοίκηση, οπότε μιλάμε για ένα one-stop shop. Σημαντική πτυχή είναι πως μπορεί έτσι να ενοποιήσει κέρδη και ζημίες, σημαντικό αυτό για την εσωτερική αγορά. Σημαντικό επίσης πως ε, τα κέρδη τα οποία ε, γίνονται εδώ πέρα να μοιραστούν σε όλα τα κράτη-μέλη στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία με βάση μια κλίδα που έχει τρεις ε, παράγοντες, δηλαδή την εργασία, τα ενεργητικά και τις, πράξεις και βεβαίως το κόστος είναι όπως είπαμε το εργασιακό και τα παγιακόστη και βεβαίως ε, θα πρέπει, όπως είπαμε, να υπολογιστεί αυτή η φορολογική βάση και θα γίνεται ένας υπολογισμός αυτής της φορολογικής βάσης και θα μπορεί να κατανέμεται σε όλα τα κράτη-μέλη και μετά επαφίεται στο κάθε κράτος μέλος ελεύθερα να ορίσει ποιο θα είναι το ύψος της φορολογικής κλίμακας και βεβαίως θα μπορεί μετά να ορίσει και αν θα υπάρχει διαφορετική κλίμακα για την επιχείρηση η οποία θα δραστηριοποιείται με την κοινή ενωπημένη φορολογική βάση και για αυτές οι οποίες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο εθνικό πλαίσιο. Και μετά υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί, διαδικαστικοί κανόνες, προβλέπουμε να μην υπάρξει κατάχρηση, αυτό βέβαια σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε Υπάρχουν επίσης ε, ζητήματα τα οποία προβλέπονται να πάνε κάτω εξοδότηση και κάτι το οποίο είναι σημαντικό πως προβλέπεται και ένας πίνακας αντιστοιχίας με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα λοιπόν περιορίζεται πολύ απλά να σας το πω το ε, διοικητικό κόστος, η ενοποίηση επίσης των λογιστικών καταστάσεων είναι κάτι το πολύ απλό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ενοποίηση, όπως είπα, ζημιών και κερδών. Αποφεύγουμε τη διπλή φορολόγηση, για το οποίο υπάρχουν κανόνες στην Ευρώπη. Γιατί παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει διπλή φορολόγηση, αποκλείεται πλέον με αυτό το σύστημα. Επίσης, τελειώνει τελειώνουν ε, κάποια προβλήματα όπως το transfer pricing που ε, ορίζουμε πλέον το τι επιτρέπεται, το τι δεν επιτρέπεται. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις με τις διοικήσεις και είχαμε ε, προβλήματα, ξέρετε, με τις διοικήσεις, με τις επιχειρήσεις και κατέληγαν με την εφορία στα δικαστήρια και αυτό λοιπόν τελειώνει. Επίσης γίνονται πολύ πιο πρακτικά και απλά το να διαρθρωθεί μια επιχείρηση και να συνεχίσει να λειτουργεί διασυνοριακά, όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται σε μια εσωτερική αγορά. Επίσης γίνεται πολύ πιο διάφανο το σύστημα, δηλαδή θα έχουμε μια κοινή δήλωση κατ' ουσίαν έναν ισολογισμό ο οποίος θα είναι πανευρωπαϊκός και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί θα είναι κοινοί οι κανόνες και βεβαίως μπορούμε να παρατηρήσουμε μετά πως καμιά φορά γίνεται λόγος για την πρόταση αυτή και εδώ μέσα και εκτός ως εάν να επρόκειτο για μια βάση για τα ίδια μέσα της κοινότητας στο μέλλον, στο απότερο μέλλον θέλω να σας καθησυχάσω, δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, ε, απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα γίνει πιθανώς στο απότερο μέλλον, αλλά δεν το συζητάμε τώρα το υπέρ ή κατά αυτού του στήματος είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει άλλη φορά. Οπότε, απλά πρέπει ε, δεν ξέρω. Ε, επίσης ε, για αυτό το οποίο ακούστηκε πως πάμε προς μια εναρμόνιση των κλιμάκων των φορολογικών και σε αυτό να σας καθησυχάσω τα κράτη διατηρούν την φορολογική τους κυριαρχία και την ανεξαρτησία σε αυτό. Βεβαίω δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα και είναι ευχαρίστηση για το ότι είμαι εγώ εισηγήτρια για κάτι το οποίο ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πάνω από 10 χρόνια. Πραγματικά αναγκάστηκα να κοιτάξω 10 χρόνια στο παρελθόν. Μπορώ να περιοριστώ όμως μόνο στο τωρινό ημερολογιακό έτος. Μόνο φέτος είχαμε τέσσερα ψηφίσματα με τα οποία ζητούσαμε την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση τον Απρίλιο, το Μάιο στο ψήφισμα για το Small Business Act που λέμε πως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξυπηρετηθούν από την εσωτερική αγορά καλύτερα. Επίσης το συζητήσαμε στο ψήφισμα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης το αναφέραμε τον Ιούλιο όταν ψηφίσαμε το ψήφισμά μας για την κρίση όπου πάλι αναφέραμε την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για ένα μέσο καταπολέμησης της κρίσης. Το είχαμε συζητήσει και το 2010, με την έκθεση Μπερσάνη, 2005, συγκεκριμένη έκθεση για αυτό το θέμα, με βάση ένα non-paper της ε, Κομισιόν και βεβαίως νομίζω πως ε, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αφετηρία μιας έκθεσης και Βλέπετε, το ήταν κάτι το οποίο ζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Η Επιτροπή μας μαζί με τους ειδικού από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν εργάστηκε χρόνια για να, καταλήξει σε, για να καταλήξει σε αυτή την πρόταση και νομίζω πως τελικά είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, μια πάρα πολύ καλή βάση συζήτησης, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε. Συγκεκριμένα τώρα για την ε, έκθεση αυτή νομική βάση είναι το άρθρο 115, άμεση φόρη, το οποίο απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών και εμείς έχουμε μόνο μία, έναν συμβουλευτικό ρόλο. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε το Συμβούλιο Υπουργών. Αυτό δεν θα γίνει βεβαίως να ασχοληθούμε με όλες τις λεπτομέρειες, το τι εκπίπτει και το τι όχι από όλα τα άρθρα θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια για να γίνουν α, αυτές οι αλλαγές ε, στα κράτη μας τα ίδια έτσι ώστε η αλλαγή η οποία θα προκύψει στο τέλος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη έτσι ώστε το κόστος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις μας να είναι μικρότερο και να μην έχουμε μετά τόσο πολλά προβλήματα. Και έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή και βεβαίως αν έχουμε ευρεία πλειοψηφία θα μπορούμε να σταθούμε σε, κάποιες, σε κάποια κρίσιμα πολιτικά σημεία. Και ένα τέτοιο σημείο είναι πρώτα απ' όλα όπως είπα ο χαρακτήρας ο οποίος είναι προαιρετικός. Τι άποψη έχουμε εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών. Το είχαμε ζητήσει στην έκθεση αυτό ήταν το 2005, εντωμεταξύ είμαστε στο 2011 και αν τεθεί ενισχύ η κοινή φορολογική βάση, μιλάμε για το 2013, Τελείω διαφορετική εποχή. Οπότε το ερώτημα το πρώτο είναι εμείς ως Κοινοβούλιο εξακολουθούμε να είμαστε υπέρ του προαιρετικού χαρακτήρα ή όπως το πιο πρόσφατο ψήφισμα μας είμαστε υπέρ του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Ε, πρέπει να τοποθετηθούμε ω προς αυτό. Υπάρχουν υπέρ και κατά και για τις δύο απόψεις. Ε, ο χαρακτήρας ο προαιρετικός μας δίνει τη δυνατότητα μιας πιλωτικής φάσης. Επίσης έχει το πλεονέκτημα το ότι μπορεί να ε, επιλεγεί από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μία χώρα αλλά έχουν διεθνείς φιλοδοξίες αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι κάποια πλεονεκτήματα. Επίσης σεβόμαστε την κυριαρχία των κρατών μελών αλλά μειονέκτημα είναι το ότι αν είναι κάτι το οποίο είναι κάτω επιλογή είναι πως όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, τα οικονομικά τα οποία αναφέραμε θα περιοριστούν βεβαίως. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν σκιώδη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Και βεβαίως το εάν μπορέσουμε να ελοπίσουμε ένα τέτοιο σύστημα για 27 κρατημέλη ή θεωρούμε πως πρέπει να ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσει δηλαδή αμέσως η κάθε χώρα να ξεκινήσουν πρώτα απ' όλα στην Ευρωζώνη ας πούμε ή με μια συνεργασία των όσων θέλουν χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα την Ευρωζώνη. Και βέβαια μπορεί κάποιο κράτος να αλλάξει μετά γνώμη. Στην έκθεση του 2005 μίλησαν για μια στενή συνεργασία. Ίσως κάποιοι να θεωρούν πως αυτό αρκεί. Τώρα, ενοποίηση κερδών και ε, πολιών και ζημιών εάν δεν ε, προβλέψουμε κάτι τέτοιο από ό,τι μου λένε όλοι δεν έχει τότε κανένα νόημα γιατί εάν δεν προβλεφθεί κάτι τέτοιο τότε κατ' ουσίαν δεν ε, κάνουμε τίποτα. Για το One Stop Shop βεβαίως δεν φαντάζομαι να είναι κανείς κατά σε κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά βέβαια στις διοικήσεις, οι οποίες κανονικά υπηρετούν την πραγματική οικονομία και νομίζω πως το σύστημα αυτό του One Stop Shop είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε μια διοικητική απλοποίηση μέσω βεβαίως ε, και των απαραίτητων εφαρμοστικών μέτρων. Τώρα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δεν ε, προχώρησα εγώ σε υπολογισμό, αλλά διάβασα κάποιες εκθέσεις. Θα γίνει ευρύτερη λοιπόν η φορολογική βάση, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από το ότι θα έχουμε, όπως είπα, ενοποίηση κέρδους και ζημιών. Χωρίς να μειωθεί να μειωθούν τα έσοδα των κρατών μελών πρώτων αυτών. Δεύτερον, υπάρχει μια ευρεία βάση και αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη που το θέλουν να μειώσουν τον φορολογικό συντελεστή για να είναι αυτή η πρόταση φορολογικά ουδέτερη. Κατόπιν έχουμε, όπως είπα, τον συντελεστή που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ειδικά εφόσον μιλάμε για άμεσους φόρους, το έχουμε πει αυτό το πράγμα ερετός, αλλά στο τελευταίο ψήφισμα ζητάμε να υπάρχει ένα όριο ανώτατο και κατώτατο. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ κάτι τέτοιο, νομίζω πως θα είναι ένα άλμα, είμαστε σε περίοδο κρίσης, θα πρέπει να πούμε το τι θέλουμε και το ποιο θα ήταν για εμάς το ιδεώδες, από την άλλη βεβαίως αν είμαστε ρεαλιστές πρέπει να παραδεχτούμε πως τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν ένα τέτοιο βήμα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε, να μάθουμε κάτι και να κάνουμε μία απόπειρα να καταλήξουμε σε μία θέση κατόπιν. Θέλω να τονίσω πως την πρόταση αναφέρεται, πως αυτό είναι και παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών για να μην μπλέξουμε τώρα. Και Κάποιοι λένε πως πρέπει να οδηγηθούμε σε ε, ενιαίο συντελεστή, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε φορολογικό ανταγωνισμό. Κοιτάξτε, φυσικό είναι να έχουμε φορολογικό ανταγωνισμό και θα ήταν πολύ πιο απλό και διαφανές να έχουμε έναν ενιαίο συντελεστή. Και ο φορολογικός ανταγωνισμός δεν είναι κάτι το κακό επίσης, έχει τα πλεονεκτήματά του. Αρκεί ε, βεβαίω να μην βλάπτει τον στόχο που έχουμε ως ευρωπαϊκή αγορά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Για το εάν θα πρέπει, όπως είπα, να έχουμε μια ψαλίδα εντός της οποίας θα κινούνται τα, τα αυτά. Η κλίδα, ο τύπος κατανομής μεταξύ των κρατών μελών που ανησυχεί τον κόσμο, τα τρία αυτά κριτήρια. Εγώ θεωρώ πως δεν είναι τίποτα το καινούριο αυτό το κριτήριο, είναι δοκιμασμένο ήδη. Ε, έχουν υπάρξει παρόμοιες αποφάσεις. Επίσης ε, συζήτησα με την Κομισιόν και τους πιστεύω πως ε, αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων εδώ και καιρό και είναι αυτό το οποίο προσφέρεται λιγότερο για καταχρήσεις. Επίσης, ρήτρα για την αποφυγή καταχρήσεων μας λένε πλέον πως πρέπει να έχουμε ειδικέ ρήτρε για την αποφυγή καταρτήσεων, αλλά εδώ πέρα ξεκινάμε με ένα νέο σύστημα και νομίζω πως καλό είναι να έχουμε μια γενική ρήτρα και μετά το ειδικό, το συγκεκριμένο μπορεί να προκύψει όταν θα έχουμε και εμπειρία. Ε, κατόπιν έχουμε τέσσερα θέματα όπου η Κομισιόν προτείνει να πάνε σε πράξεις ε, κάτω εξουσιοδότηση και να δοθεί αυτή η εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως θα έχουμε και τον πίνακα αντιστοιχίας. Αυτό νομίζω είναι προφανές, δεν χρειάζεται εξήγηση. Οπότε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Γιατί εκεί πέρα αναμένουμε, εκεί πέρα πρέπει να αναμένουμε γιατί ε, απαιτείται ομοφωνία. Οπότε, ένα άλλο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν να μην συμπίπτουν αυτοί οι κανόνες με τους λογιστικούς κανόνες της Ευρώπης. γιατί ε, όπως έχω μάθει εγώ στο παρελθόν όσο πιο πολύ κοντά είναι αυτά τα πράγματα τόσο λιγότερος χώρος ε, δημιουργείται τον οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό στην Κομισιόν και τρίτο ερώτημα το ερώτημα για το αποτέλεσμα που θα έχει σε περιφερειακές και τοπικές αρχές η πρόταση αυτή κάποια κράτη-μέλη είναι ομοσπονδιακά αλλά έχουν περιφέρειες με φορολογική αυτονομία που μπορούν δηλαδή να επιβάλλουν φόρους σε εταιρείε. Υπάρχουν διάφοροι ε, φόροι Κοιτάξτε, για εμένα είναι σαφές. Κάνουμε κανόνες για 27 κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη μετά θα το μεταφράσουν στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές. Δεν βλέπω το πρόβλημα, αλλά κάνει κάποιους θορύβους η Επιτροπή των Περιφερειών και θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας ενημερώσει και να σχηματίσουμε και γνώμη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τους ε, συναδέλφους και βεβαίως είμαι διατεθειμένη ανά πάσα στιγμή της ημέρας ε, να δούμε ε, το ζητήμα του συναδέλφου για να έχουμε όσο δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την περιεκτική εισαγωγή. Έχουμε λίγο χρόνο, θα πάρουμε τους κοιόδη. Στις 29 Νοεμβρίου θα έχουμε την παρουσία τη έκθεση. Αν χρειαστεί μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος ε, για να εκφραστούν οι απόψεις. και ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Λίζα Φερέρα πρώτη από τους σοσιαλιστές παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ε, χαιρετίζοντα προσωπικά αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και την θετική τοποθέτηση από πλευράς της κυρίας ε, Τάισεν για αυτό το θέμα που εμείς πραγματικά εργαστήκαμε γι' αυτό και επ' αυτού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να δώσουμε ένα, να υπάρξει αυτό το θετικό μήνυμα και που θα δώσει κίνητρα να υπάρξει συνέχεια σε μια ενεργηγό τοποθέτηση από το Ευρωκοινοβούλιο που θα οδηγήσει το Συμβούλιο να αποφασίσει, να λάβει απόφαση τελικά για αυτό το θέμα. Όμως ζήτησα να παρέμβω όχι προσωπικά, αλλά εξ του συναδέλφου Λίμα Νιόκ που είναι σκιώδης εισηγητής και που για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να παραστεί ζητεί συγγνώμη και έχει ένα κείμενο το οποίο μου ζήτησε να σας διαβάσω. Θα σας διαβάσω το κείμενο που ακολουθεί και είναι το κείμενο του συναδέφου Σκιώδου εισηγητού που εξ ονόματος του PSD της ε, ομάδας των Σοσιαδημοκρατών θέλει να, να διαβαστεί το κείμενο, δεν μπορεί να παραστεί. Πολλά από τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί ε, αναφέρονται υπάρχει μια πρώτη προσπάθεια να απαντηθούν. Σας διαβάζω λοιπόν το κείμενο. Καλωσορίζω την ιδέα του CCTB. Είναι πρώτο βήμα για τον φορολογικό εναρμονισμό. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι επαρκώς φιλόδοξη. Ο μόνο, το μόνο κίνητρο για αυτό το ε, κείμενο είναι να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και να εξοικονομηθούν πόροι ούτε γίνεται λόγος για την ανάγκη καταπολέμησης του φορολογικού dumping και της υπονόμευσης των δημόσιων οικονομικών όσον αφορά τον ανταγωνισμό προς τα κάτω για την φορολογική εξυπηρέτηση. Πρέπει να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση για τη φορολογία επιχειρήσεων και φορολογία εργασίας και να υπάρξει βελτίωση των ελέγχων ε, ε, φορολογικών ελέγχων θα πρέπει εδώ να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις επιχειρήσεις και θα πρέπει η βάση αυτή να χρησιμοποιείται για να καταπολεμηθεί το dumping, το φορολογικό dumping. Όμως όπως έχει η πρόταση της Επιτροπής έχει πολλές ελλείψεις. Πρώτον, το CCCTB είναι μόνο εθελοντικό, σε εθελοντικό πλαίσιο. Και εδώ λοιπόν κάθε εταιρεία η ίδια θα είχε την επιλογή να προσυπογράψει ή όχι και να συνεργαστεί μέσα στο πλαίσιο του νέου συστήματος, ανάλογα με το τι θα ήταν πιο επωφελές. Το μείζον επιχείρημα της Επιτροπής είναι να δικαιολογήσει τον εθελούσιο εθελοντικό χαρακτήρα λέγοντας ότι δικαιολογείται αυτό επειδή μόνο κάποιες εταιρείες έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες και συναλλαγές. Αυτό το επιχείρημα όμως είναι βάσιμο όταν έχουμε το θέμα της παγίωσης, consolidation. Όταν βλέπουμε ότι διαφορετικές εταιρείες δρούν σε διάφορα κράτη-μέλη, αυτό δεν παρακολεί το να υπάρξει μια κοινή βάση προτείνω ένα, ένα εναλλακτικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δίνει προτεραιότητα, δίνει στα συμφέροντα των εταιριών εις βάρος της φορολογικής δικαιοσύνης. Όπως αναγνωρίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις του CCCTB στα έσοδα τα φορολογικά των κρατών θα εξαρτηθεί από στρατηγικές επιλογές που θα γίνουν ζητείται από τα κράτη-μέλη να αναλύσουν την κατάσταση, να δουν τι θα γίνει. Ένα άλλο πρόβλημα που απορρέει από την πρόταση CCCTB είναι ότι θα ήταν ευνοϊκή ρύθμιση μόνο για τις πολυεθνικές ε, εταιρείες. Μόνο μια μειονότητα μικρών εταιρεών δρούν σε περισσότερα κράτη-μέλη και δεν έχουν τις δυνατότητες να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα. Γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος οι μεγάλες εταιρείες να επιλέξουν το CCCTB και να ελαφρυνθεί, να διευκολυνθεί το φορολογικό τους βάρος σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο όχι μόνο δεν είναι δίκαιο, αλλά θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις και για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με τον εθελοντικό χαρακτήρα του CCCTB, το βάρος θα μετατίθεται από οι επιχειρήσεις που δρούν στα κράτη-μέλη σε ε, άλλα στα συστήματα των εθνικών κρατών και το CCCTB. Η πρότασή μου, η πρόταση του Λίμαν λοιπόν, από πλευράς Λίμαν είναι η εξής. Το πρώτο είναι φυσικά ότι η βάση, η κοινή βάση αυτού του κειμένου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικού, δεσμευτικού χαρακτήρα. Δεύτερον, η παγίωση δεν πρέπει να οδηγήσει ως consolidation σε ακραίες περιπτώσεις μη φορολόγησης ή άδικη φορολόγηση. Για παράδειγμα, με ένα ελάχιστο κατόφλι φορολόγηση που θα πρέπει να καλύπτεται από μια εταιρεία για να υποφελείται αυτή από το CCCTB. Εδώ μπορούμε να εμπνευστούμε από αυτά που προτάθηκαν πρόσφατα στην έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ για τους κανόνες που θα ισχύουν για μητρικές επιχειρήσεις και θυγατρικές επιχειρήσεις. Εν τέλει το CCCTB θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συντονισμό ή ένα αρμονισμό των ποσοστών. Η πρότασή μου θα ήταν να υπάρξει μια δυνατότητα ευρωπαϊκής φορολόγησης όσον αφορά και το ότι ίσχυε στο παρελθόν όταν είχαμε διαφορετικά νομίσματα. Θα θέλαμε να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ της φορολόγησης των κρατών μελών και να αποφύγουμε στρεβλώσεις. Σαν ένα πρώτο βήμα λοιπόν για τα θέματα τα οποία αναφέρονται εδώ Κάποια από αυτά απαντώνται, την χάνουν απαντήσεων από πλευράς Λίμαν. Θα έχουμε όμως ευκαιρίες να ανταλλάξουμε απόψεις από αυτών των θεμάτων υστερότερα και να καταλήξουμε σε μια συντονισμένη κοινή θέση για το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την Άλντε. Έχετε εσείς τον λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ τη Μαριάν για την πολύ πλήρη αυτή παρουσίαση. Δεν θέλω να επισέλθω καθόλου σε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή, γιατί συμφωνώ απόλυτα ένα πρώτο ζήτημα το οποίο τίθεται και το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου για το άρθρο 115 και την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Μπορούμε να επανεφεύρουμε ό,τι θέλουμε, αν μας ευχαριστεί αυτό, αλλά ίσως εισακουστούμε, αν εισακουστούμε, αν είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς σε κάτι που είναι πολιτικά ξεκάθαρο και λογικό. Δεύτερον, έχουμε το πλαίσιο της κρίσης και όλες οι προτάσεις ε, που είναι στα σπάργανα ακόμη και δεν τις έχουμε ακόμη ξεκάθαρες ε, και όπως, είπε και ο, όπως ξέρει και ο Τιώγο Φέιο έχουμε ένα ε, σχέδιο το οποίο έγινε πριν, όχι προ Χριστού, νωρίτερα όμως, 10 χρόνια πριν, έχουν γίνει μικρά βήματα. Άρα Λίγο αντιφατικέ οι δύο παρατηρήσει. Πρώτο, θα μπορούσαμε να δεχθούμε αυτό που προτείνει η Κομισιόν, λέγοντα ότι τελικά είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά το επιχείρημα τη εσωτερική αγορά, με πείθει ιδιαίτερα, που ξέρουμε ότι δεν τα πάει και πολύ καλά η εσωτερική αγορά. Απ' την άλλη πλευρά όμω, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη την κρίση και το τι μπορεί αυτή να σημαίνει, γιατί θέλησε να πάμε πιο πέρα, ιδίω ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα αντίθετα συμπεράσματα. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν έχω καταλήξει. Νομίζω ότι καλό είναι να μιλήσουμε όλοι, να ακούσουμε ένα τον άλλο και να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα της ενοποίησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και ορθό. Καταλαβαίνω ότι πράγματι ευνοούνται οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι προφανές όμως ότι προσπαθούμε να έχουμε ένα 28ο καθεστώς μέσα στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι ο στόχος. Όχι να έχουμε την τοπική άσκηση δραστηριοτήτων από τι επιχειρήσει. Η τάση μου είναι να προτιμώ να δράσουμε σε επίπεδο 27. Όχι αποκλειστικά, όχι με αποκλειστικό τρόπο, να δούμε δηλαδή τι μπορεί να θέλουν οι υπόλοιποι και να διατηρήσουμε σίγουρα την εσωτερική αγορά των 27. Απ' την άλλη όμως, όσοι δεν θέλουν τίποτα, δεν θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να μπλοκάρουν τους υπόλοιπους. Από τη στιγμή που προσπαθήσαμε και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, βέτο κτλ, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ενδεχομένω κάποιες άλλε μορφές ε, κάποιες άλλες οδούς, ίσως ενδεχομένως ενισχυμένη συνεργασία. Όλα πρέπει να μείνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Σταματώ εδώ, αλλά ετέθη και το ζήτημα αυτό της ε, κλίδας, ε, ενεργητικό, ε, τζίρος, εργασία, αγορά εργασίας. Δεν ξέρω ακριβώς τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την κρίση πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας σε σχέση και με αυτή την κλίδα. Λοιπόν, χαίρομαι που ε, η Μαριάννα έχει κάνει μια πολύ καλή πρώτη απόπειρα. Θα συνεργαστούμε μαζί της και ελπίζω με ευφύ τρόπο και με τους υπόλοιπους. Σίγουρα η φορολογία είναι στο επίκεντρο του δημοκρατικού διαλόγου. Και είναι ένα θέμα που, ας μην αυτοπαθούμε, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και στο μέλλον. Από το ECR ο κύριος Στρέτσεκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα την κυρία Τίσεν με πολύ μεγάλη προσοχή. πραγματικά περίμενα με ανυπομονησία να δω πώς θα ξεφύγει, πώς θα ξεπεράσει το ότι ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο μπορούν να εναρμονίσουν ε, την άμεση φορολογία. Μάλλον θα είμαι ένας μοναχικός καβαλάρης στην Επιτροπή. Το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Θα προσπαθήσω πάντως να προσπίσω τη δική μου θέση. Την οποία θεωρώ σημαντική και κρίσιμο. Καταλαβαίνω. Το ανέφερε αρκετές φορές και η κυρία Τίσεν. Καταλαβαίνω την προσπάθεια που επιχειρείται να γίνει κάτι με μια διαδικασία που θα ολοκληρώσει τη φορολογική ένωση χωρίς όμως να ακουμπήσει τους άμεσους φόρους. Αλλά χωρίς την άμεση φορολογία είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Άρα κάτι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η φορολογική ένωση. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτό είναι αδύνατο να γίνει με συντελεστέ. Το είπατε, το είπατε πολλές φορές. Εξού και υπάρχει μια πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιριών. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο φόρος, ε, η φορολόγηση είναι μια διαδικασία όπου η φορολογική βάση πολλαπλασιάζεται επί το φορολογικό συντελεστή, τον εκάστοτε. Τώρα δεν ξέρω ποιο μέρο τη διαδικασία μπορεί κανεί να προσπαθήσει να αναρμονίσει και δεν έχει και σημασία. Τελικά το ίδιο αποτέλεσμα θα προκύψει. Οι φορολογικοί συντελεστέ δεν είναι πλέον σημαντικοί. Η φορολογική βάση όμω είναι σημαντική. Και πρόκειται για μια προφανή απόπειρα εναρμόνισης των άμεσων φόρων από την πίσω πόρτα, αν με επιτρέπει η έκφραση. Πρέπει να το πει κανείς. Και καλό είναι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματά σας και τη θέση σας. Καταλαβαίνω και κατανοώ τη θέση, φαντάζομαι, και των υπολείπων. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι μια απόπειρα να γίνει κάτι με την άμεση φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν θέλω να μιλήσω για κόκκινες γραμμές ή κάτι τέτοιο. Φυσικά και είμαι διατεθειμένος και πρόθυμος να συνεργαστώ και να συνεργαστώ μαζί σας αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που μου φαίνονται ουσιώδη. Είναι θέματα αρχής για μένα. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι λέτε ότι θα είναι αυστηρά προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό αυτό το σύστημα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο με βοηθά να μπορέσω να συνεργαστώ, να είμαι συνεργάσιμος. Τώρα, σε αυτό το σύστημα του CCTB, τη κοινή ενωπημένη βάση δραστηριότητα των εταιριών, αυτό ίσω να είναι αποτέλεσμα διακυβερνητική συμφωνία. Συμφωνία διακυβερνητική μεταξύ των κρατών μελών. Στην προκειμένη περίπτωση, και αν το κάνουν οι χώρε, αυτό δεν έχω πρόβλημα. Πάντω, είμαι κάπω δύσπιστο. Αν αυτό το σύστημα εισαχθεί ως ένα σύστημα παράλληλο με τα εθνικά συστήματα. Μήπως αυτό αυξήσει το διοικητικό κόστος και αθέλητα, και το τονίζω αυτό, αθέλητα αυξήσει και το διοικητικό άχθος. Επίσης, η ενοποίηση, και τονίζω τη λέξη αυτή, η ενοποίηση θα αντισταθμίσει τις απώλειες οι οποίες θα προκύψουν από την ανακατανομή του πλούτου. Από τις θηγατρικές ή Και είναι θέματα που μπορεί, ε, για τα οποία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εσύ εξ ονόματος των Πρασίνων, γιατί είχα Λάμπερτ, δυστυχώς ο Φίλιπ δεν μπορεί να παραστεί, είναι σκιώδης. Έτσι εγώ θα τοποθετηθώ γι' αυτόν. Όπως πάντα βρισκόμαστε όμως πολύ κοντά στις απόψεις μας ο ένας ε, με τον άλλον. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη αφορά την πολιτική και εσείς ε, διαρωτάστε ποιες χώρες μπορούν να τα καταφέρουν και να το κάνουν σε σχέση με την δυνατότητα να λειτουργήσει αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταφέρουμε. Προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόταση θα ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη. Κάποιες χώρες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις. Παράλληλα έχουμε και την διεργασία του Europlus Pack. Υπό αυτή την πρόταση τουλάχιστον 23 κράτη-μέλη υπέγραψαν ότι θα κινούνται προς ένα τέτοιο σύστημα και τέσσερις ε, χώρες για διάφορους λόγους δεν εντάχθηκαν σε αυτές τις άλλες 23. Ενδιαφέρον ήταν να δει κανείς στην απόφαση μείωση των επιτοκίων για την υποστήριξη του προγράμματος χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την παγιωμένη φορολόγηση επιχειρήσεων ενιαία, σε ενιαία βάση. Θα τα δω πολύ προσεκτικά, θα τα παρακολουθήσω αυτά, αλλά έχοντας ακούσει για τις δύο διαφορετικές ομάδες που έχουν μια συγγενή σύνθεση η μία είναι εκείνη που προσεγγίζει το Συμβούλιο, η άλλη εκείνη που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Φορολογία Επιχειρήσεων. Όμως ε, δεν είναι ακόμα επικοδομητικό το πλαίσιο. Έχουμε την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία. Ακούω ότι υπάρχει κάπως πιο προσεκτική αντιμετώπιση σε σχέση με το Βέλγιο όσον αφορά το παρελθόν. Όμως χρειαζόμαστε ομοφωνία και αν δεν υπάρξει αυτή μπορεί να τροχοπεδηθεί η πρόοδος. Όπως γνωρίζετε υπάρχει η Γερμανογαλλική Σύνοδος Κορυφής που αποφάσισε να κινηθεί προς ένα κοινό γαλλογερμανικό σύστημα φορολόγησης εταιριών που θα είναι πιο ισχυρό ακόμα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε απόλυτα τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο μεγαλύτερες χώρες μέλη λένε «Προσέξτε, εφόσον υπάρχει θέμα με τις μικρότερες χώρες για να γίνει κάτι συνετό, διότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να υποφεληθούν από την μετάθεση ε, φορολόγησης, θα δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ζώνη και θα υπάρξει πίεση. Γιατί εδώ σε σχέση με τις εταιρείε που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται στην Ευρωζώνη, και που θα πρέπει με διαφορετικά συστήματα φορολόγησης ε, να ε, αντιμετωπίσουν, δεν επιθυμούν να αντιμετωπίσουν το κόστος ε, σε σχέση με τα διαφορετικά κράτη-μέλη και ο καθένας να προσπαθεί από πλευράς της κοινή βάσης φορολόγησης να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η στάση τροχοπέδησης οδηγεί τώρα στο να προσεγγίσουμε μια μη κοινοτική βάση εναρμονισμού. Πράγμα το οποίο ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να επιθυμούμε με κανένα τρόπο, διότι όπως είναι αποδυναμωμένες οι εξουσίες μας ήδη επ' αυτών των θεμάτων σήμερα, αν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πιο αποδυναμωμένες οι αρμοδιότητές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της νομικής βάσης, αλλά να προσπαθήσουμε στα εκτιμώντα τι αιτιολογικές ε, σκέψεις να αντιμετωπίσουμε το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ένα δεύτερο σημείο παρατήρηση που θα ήθελα να αναφέρω επίσης είναι ότι Όλη αυτή η συζήτηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό για μένα ξεπερνά τα τεχνικά θέματα. Είναι φιλοσοφική υφής συζήτηση. Η ιδέα της επικουρικότητας, όπως αναφέρεται στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέρχεται από την ηθική της κοινωνικής ε, συμβίωσης, η ιδέα όχι του να απέχει κανείς από κάποια πράγματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να τα κάνει όλα στο χαμηλότερο επίπεδο όπου μπορεί να υπάρχει έλεγχος και να μπορεί να υπάρχει και ε, κυριαρχία. Όμως στην φορολογία δεν υπάρχει εθνική ε, κυριότητα, εθνική κυριαρχία. Μπορούμε να έχουμε κανόνες και κανονισμούς, όμως μπορεί να ε, υπεκφεύγουν κάποιοι με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν καθιστούν εφικτή την χρήση του, της εθνικής κυριαρχίας. Και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε και να μην δημιουργούμε σύγχυση. Και όταν αναφέρονται σε κυριαρχικά δικαιώματα κάποιοι, αυτό που θέλουν είναι να προασπίσουν πλεονεκτήματα και <clears throat> προνόμια κάποιων εταιριών για την κατάχρηση όσον αφορά τις ε, διατάξεις για την ε, φορολογία. Ενώ επιχειρήσεις που δεν το κάνουν αυτό, που πληρώνουν τους φόρους τους ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δυνατότητα υπεκφυγής επειδή δεν είναι πολυεθνικές και είναι μικρές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν αθέμητο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά, όπου υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να κάνουν κατάχρηση των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων και άλλες που ή για ηθικούς λόγους δεν θέλουν να το κάνουν ή δεν μπορούν ε, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν εδώ για παράδειγμα πολύ την ε, δραστηριοποίησή τους σε ένα επίπεδο που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους ε, αποφυγή φορολόγησης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την ε, πίεση που θα μπορέσει να δημιουργηθεί έναντι των κρατών μελών για την, να κινηθούν προς χαμηλότερα ποσοστά φορολόγησης. Θα υπάρξει ανταγωνισμός αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρύθμιση. Γι' αυτό πρέπει να προβούμε σε μια ε, σε έναν εναρμονισμό της, βύση, της βάσης. Πρέπει να υπάρχει και ένας, ένας ελάχιστος εναρμονισμός, ε, συντονισμός της φορολογικής βάσης. Και όπως είπαμε σε σχέση με το πλαίσιο για τη δική μου έκθεση που δεν ε, χρειάζεται να ε, απαγορεύεται, να, να απαγορεύει ε, γιατί δεν θα αποκλείται από ένα κράτος να, ε, να πάει προς τα εμπρός αλλά η ίδια η πραγματικότητα θα δημιουργεί φραγμούς και όρια. Και πιστεύω δεύτερον θα πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα αυτές οι ρυθμίσεις. Αν δεν είναι δεσμευτικές αυτές οι ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες περιπλοκές. Θα πρέπει τουλάχιστον να είναι δεσμευτικές για τις μεγαλύτερες εταιρείε. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε το πρόβλημα διαρκώς της σύγκρισης διαφορετικών φορολογικών συστημάτων, πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και επιβάρυνση και θα είναι πολύ περίπλοκο το θέμα των επιλογών του πώς να καταφέρει κανείς να πληρώσει λιγότερους φόρους στο τέλος τέλος. Και εν τέλει υπάρχουν κάποιες χώρες που φοβούνται για την φορολογική τους βάση και ανησυχούν και επειδή έχουν προβλήματα ίσως θα μπορούσε να υπάρξει ένας νέος, ε, ε, μιας νέας μορφής ε, υπονομευτικής θετικός ανταγωνισμός ε, όσον αφορά την ε, φορολόγηση, ανταγωνισμός ε, dumping προς τα κάτω. Θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανονισμοί και η αποτελεσματική εποπτεία, γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτά είναι οι πρώτες ιδέες ως στοιχεία σημαντικά για αυτές τις προτάσεις και η πραγματικότητα έλλειψης ρευστού σε σχέση με τα διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρώπης θα βοηθήσει ίσως να επιληθούν κάποιες από τι ιδεολογικέ διαφορές που έχουμε και που αντιμετωπίζει προβλήματα και το Συμβούλιο και θα ελπίζουμε ότι θα κινητοποιηθούν τα πράγματα αν δούμε τι γίνεται σε σχέση με τη ρευστότητα των κρατών μελών σήμερα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Εγώ ήθελα ρωτήσω κάτι την Κομισιόν. Βεβαίω δεν υπάρχει χρόνο για συζήτηση. Θα ήθελα να μάθω εάν προχωρήσει η ομάδα Europlus, ας πούμε, ή μια πιο περιορισμένη ομάδα με αυτή την πρόταση. Είναι κάτι το ενδιαφέρον το οποίο μπορούμε να, κάτι το οποίο μπορείτε να κοιτάξετε. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις εταιρείες εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να αποφεληθούν από μια πανευρωπαϊκή κοινή φορολογική βάση. Καταλαβαίνω ότι τα πλεονεκτήματα να το κάνει κανείς. Εάν είναι απ' έξω κάποιο θα υποφέρουν οι εταιρείε. Δεν περιμένω να το απαντήσετε τώρα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα για εμένα συζήτηση, καθώς γίνεται στα κράτη-μέλη που έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στο σύστημα. Και δεν μιλάω μόνο για την γραφειοκρατία. Οπότε είστε διατεθειμένοι να κοιτάξετε κάτι τέτοιο. Και μετά θα δώσω τον λόγο ξανά στην εισηγήτρια. Και νομίζω πως γίνεται μια άλλη συζήτηση εδώ πέρα ούτως ή άλλως πριν παρουσιάσετε την εκθέση σας. Ο κύριος Νίλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία από την πλευρά της Κομισιόν, η δυνατότητα αυτή είναι η τελευταία τότε που έχουμε. Η πρότασή μα είναι για τα 27 κράτη-μέλη. Εάν κάποια κράτη-μέλη θέλουν να ακολουθήσουν ενισχυμένη συνεργασία, νομίζω πως είναι σαφέ πως εάν το κάνει μια μικρότερη ομάδα από τι 27, μιλάω για το τι θεωρεί η Κομισιόν, για κάποιες εταιρείε που ε, δραστηριοποιούνται σε κάποιες χώρες, ε, σε χώρες που είναι εκτός του συστήματος, προφανώς θα είναι λιγότερο ελκυστικό αυτό σε σχέση με μια κοινή ενοποιημένη βάση. Γιατί βεβαίως τα πλεονεκτήματα, όπως τα είπε και η συγγήτρια, νομίζω πως μειώνονται ε, αν είναι λιγότερα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Αλλά νομίζω το θέμα είναι το πόσα κράτη-μέλη σε αυτήν την περίπτωση θα κάνουν κάτι τέτοιο και αν θέλετε και ποια. Αλλά οπωσδήποτε από τη σκοπιά της Κομισιόν αν έχουμε ενισχυμένη συνεργασία αναμένουμε ε, πως θα είναι λιγότερο ελκυστικό το σύστημα από ότι αν είναι και 27 χώρες γι' αυτό μάλιστα επιμένει η συνθήκη να είναι ε, και τα 27 κράτη-μέλη σε αυτές τις περιπτώσεις και η ενισχυμένη συνεργασία είναι τελευταία λύση. Κυρία Τάισεν, θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να τοποθετηθεί η Κομισιόν για την περιφερειακή πτυχή, γιατί φοβάμαι ότι αν δεν ξεκαθαρίσει θα δυσκολεύσει αργότερα την ε, συζήτησή μας εδώ πέρα. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά μπορούμε να τα δούμε και αργότερα. Αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους. Νομίζω πως οι ανησυχίες που ακούστηκαν ε, είναι πράγματα τα οποία όλοι συμμεριζόμαστε. Το ερώτημα είναι ποια είναι η καλύτερη διέξοδος για να έχουμε μια ευρεία στήριξη της έκθεσης στο Κοινοβούλιο και να οδηγηθούμε αποτελεσματικά στην καλύτερη δυνατή οδηγία την οποία πραγματικά χρειαζόμαστε. Χαίρομαι για το ότι ακούω το ότι συμφωνούμε πλην του κυρίου Στρέτσεκ ο οποίος πάει σε μια άλλη κατεύθυνση μπορούμε να το συζητήσουμε την άλλη φορά νομίζω νομίζω θα θα δούμε, μπορούμε να συζητήσουμε για να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας. Επίσης χαίρομαι κύριε Πρόεδρε για το ότι ε, συμφωνούμε γιατί θα έχουμε κάποια επιρροή μόνο εάν έχουμε ευρία συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μιλήσουμε με ενωμένη φωνή, αλλιώς η επιρροή μας θα είναι μηδενική. Αλλιώς πάμε να δούμε λίγη μπαλίτσα. Ή να κάνουμε τζόγινγκ ή ποδήλατο. Οπότε χαίρομαι για το ότι συμφωνούν και οι σκιοδησίτες και αναμένω την συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Πράγματι είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει ξανά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε νομίζω άλλη μια ανταλλαγή απόψεων θα εξετάσουμε στις 29 Νοεμβρίου το σχέδιο έκθεσης και η προθεσμία θα είναι κάποια στιγμή μετά για τις τροπολογίες.